και που παρακινεί σε διάπραξη ε, τέτοιων ενεργειών, μίσους. Δεν μπορούν ε, να ε, είναι πιο προσβάσιμα για όλους τα ιστοσελίδες εκείνες που ουσιαστικά υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Βγαίνουν πάνω-πάνω στις μηχανές αναζήτησης. Αυτό δεν είναι δυνατόν να το δεχθούμε. Επίσης, ε, πρέπει να παραμερίσουμε και να απομονώσουμε ε, χωρίς να φαίνεται ότι γίνεται αυτό, όπως ε, παράδειγμα ανέφερα στη Γαλλία, τι γίνεται στη πολιτική στην περιοχή του Παρισιού. Επίσης, οι συνθήκες κράτησης θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα αυτών των κρατουμένων, όπω και για όλου του άλλου κρατουμένου. Βέβαια, πρέπει αυτό να ισχύει. Υπάρχουν και άλλε τροπολογίε πολύ ενδιαφέρουσε που εμπλουτίζουν την έκθεση. Απλά μένει να προσπαθήσουμε να συντάξουμε συμβιβαστικέ τροπολογίε και το Σεπτέμβριο θα τα συστήσουμε όλα αυτά με του σκιώδει. Αυτά σε αδρέ γραμμέ. Ε, για τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Συνολικά νομίζω ήταν πολύ πλήρη σε πλούσια δουλειά που έγινε. Υπήρξαν και τροπολογίες που γύρουν και άλλα ζητήματα, ε, κάποιες ιδιαιτερότητες. Νομίζω ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε έναν ευφυή ενδιαφέροντα συμβιβασμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρασιντά. Κανονικά σκιώδεις ηγητές, ε, πρώτη κυρία Άννα Γκόμες. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ντατή, την εισηγήτριά μας δηλαδή, για την διαθεσιμότητά της, γιατί συνεργάστηκε πολύ καλά μαζί μας. Πραγματικά ήταν πολύ θετική η στάση της και νομίζω ότι μαζί με τους υπόλοιπους σκιώδεις συγητές μπορούμε να ολοκληρώσουμε επιτυχώς το έργο αυτό το γεγονός ότι έχουμε από κοινού υποβάλει πολλές τροπολογίες με τις οποίες συμφωνούμε δείχνει ότι υπάρχει σύγκληση απόψεων και ότι θα είμαστε σε θέση να περιλάβουμε διάφορες ευαισθησίες στην έκθεση αυτή, διάφορες προσεγγίσεις. Με έναν τρόπο ορθό όμως κάθε φορά. Και σεβόμενοι βέβαια το ότι θέλουμε καταρχάς να καταπολεμήσουμε την ρίζοσπαστικοποίηση, ενώ παράλληλα όμως θέλουμε να τηρήσουμε και να προστατεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Λύσω τώρα αγγλικά, γιατί έχω καταγράψει τις σκέψεις μου στα αγγλικά. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιοι τομεί στου οποίου ενδεχομένω να μην έχουμε καταλήξει ακόμα σε συμφωνία, αλλά είμαι πεπισμένη ότι θα καταφέρουμε και σε αυτού να βρούμε μια κάποια συνένεση το ζήτημα του διαχωρισμού στις φυλακές, δηλαδή να ξεχωρίσουμε τους ρίζος παστικοποιημένους, ενδεχομένως να είναι γλωσσικό λίγο το ζήτημα εδώ, αλλά η φυστάμενη παράγραφος όπως την έχουμε αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τη δική μου την ομάδα. Ξέρω ότι ε, αυτό αποτελεί μία από τις βασικές ιδέες στην έκθεση της κυρίας Ντατή, Νομίζω πάντως ότι είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε και την περαιτέρω ενσωμάτωση των ανθρώπων αυτών στο μέλλον, ακόμα και αν τους θεωρούμε σε μια πρώτη φάση ρίζοσπαστικοποιημένους. Αν εξ αρχής θεωρήσουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν καμία ελπίδα, τότε ούτε και εμείς έχουμε καμία ελπίδα όμως. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει περισσότερο να δούμε πώς θα καταφέρουμε να επανανσωματώσουμε τους ανθρώπους αυτούς στην κοινωνία. Πώς μπορούμε δηλαδή να επενδύσουμε περισσότερο σε δημόσιες πολιτικές επανένωσης, ενσωμάτωσης και όχι τόσο πολύ διαχωρισμού εντός και εκτός φυλακών. Όσον αφορά τώρα το διαδίκτυο, όπως τόνισε και η κυρία Ντατή, όντως ε, έχει συντάξει ένα τμήμα του κειμένου το οποίο είναι ιδιαίτερα πλήρε, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να πετύχουμε μια κάποια ισορροπία. Δεν μπορούμε στους παρόχους υπηρεσιών στο διαδίκτυο ή στο σελίδο να ρίχνουμε όλο το βάρος και να φέρουν αυτοί όλη την ευθύνη. γιατί ξέρουμε ότι πολλές φορές υπάρχει περιεχόμενο το οποίο προωθεί τη ρητορική μίσους ή προωθεί πολλές φορές και τη ρωσπαστικοποίηση. Δεν μπορούν όμως να φέρουν οι φορείς παροχής του διαδίκτυου όλο το βάρος της ευθύνης και νομίζω επίσης ότι θα πρέπει να αφαιρθούμε επίσης και συγκεκριμένα στάδια δικαστικών ελέγχων. Και είναι πολύ σημαντικό επίσης να δούμε τι προτείνεται στην έκθεση αυτή και το γεγονός ότι είναι πολύ λεπτή γραμμή ανάμεσα στα όσα προβλέπονται στην έκθεση αυτή και στη λογοκρισία, στην οποία δεν πρέπει να καταλήξουμε σε καμία περίπτωση. Πρέπει απλώς να έχουμε αποτελεσματικούς ελέγχους. Επίσης, νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερνόμαστε όχι απλώς σε αφηγήσεις όπω λέγεται στην έκθεση, αλλά και σε συγκεκριμένα παραδείγματα ή να προτείνουμε συγκεκριμένες πρακτικές για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης, ακόμα και στο διαδίκτυο. Και νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε λύσεις με την εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών. Και νομίζω ότι για το λόγο αυτό χρειαζόμαστε και τη χρηματοδοτική και όχι μόνο υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τρίτον, Πρέπει να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες στη δική μας την Επιτροπή για να καταφέρουμε να γεφυρώσουμε την προσέγγιση εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. Πραγματικά στον τομέα αυτό βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία διαχωριστική γραμμή ανάμεσα αυτό που συνήθως αποκαλούμε εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια. Ακόμα και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ συχνά κάνουμε αυτή τη διάκριση η οποία όμως δεν υφίσταται εν προκειμένου. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μια σφαιρική, ολιστική προσέγγιση, όπου θα χρησιμοποιούμε από κοινού όλα τα απαραίτητα μέσα, τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν να πετύχουμε το στόχο μας. Και ο στόχος μας είναι η καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης. Ορισμένε λοιπόν από τι τροπολογίε που έχουμε καταθέσει ακολουθούν αυτή την κατεύθυνση και νομίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και δυνηστικών υπηρεσιών, ε, πληροφοριών με μεταξύ των κρατών μελών είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε μέσω της ανταλλαγής αυτής πληροφοριών να οικοδομήσουμε περισσότερη εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών. Αποκλείεται ποτέ να κερδίσουμε τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας αν δεν εμπιστευόμαστε περισσότερο οι μεν τους δε. Και νομίζω θα πρέπει να συνεργαστούμε περισσότερο και με τρίτες χώρες. Δηλαδή με τους εταίρους που ήδη έχουμε στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, πολλοί εκ των οποίων βέβαια παίζουν ένα διπλό παιχνίδι, ας μην το ξεχνάμε αυτό, και προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε ακόμα και τις χώρες εκείνες οι οποίες συμβάλλουν στην αστάθεια. Ακόμα και σε χώρες όπως η Λιβύη μπορούμε να βρούμε κάποιους συνομιλητές. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε σταθερή κυβέρνηση στο εγγύς μέλλον στη Λιβύη, αλλά μπορούμε τουλάχιστον να καταφέρουμε να βρούμε κάποιους συνομιλητές και στη χώρα αυτή. Γιατί καταλαβαίνετε ότι μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ την κατάσταση. Λοιπόν, ολοκληρώνω λέγοντας ότι Θεωρώ ότι μπορούμε να συνεργαστούμε πολύ επικοδομητικά όλοι οι σκιώδεις συγητές με την εισηγήτρια και όλοι οι εμπειρογνώμονες προκειμένου να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα καλό συμβιβασμό. Ευχαριστώ πολύ. Ανά, η Σοφή Νετφέλτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ αντικαθιστώ την ε, Μαϊτέ Παγκάσα Ορτοντούα που είναι η δική μα σκιώδη συγγήτρια θα ήθελα να ξεκινήσω από ένα θέμα και εγώ έχω κάνει τροπολογία σχετικά και αυτό έχει να κάνει με την ορολογία που χρησιμοποιούμε και τη γλώσσα. Μιλάμε για ριζοσπαστικοποίηση και ξένους μαχητές, ε, πάρα πολύ επιπόλαια, αλλά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι. Όταν μιλάμε για ξένους μαχητές δεν είναι ξένοι για μας, δικοί μας είναι ε, πολίτες και η ριζοσπαστικοποίηση προτιμώ να αντικατασταθεί από τον όρο ε, βίο ε, εξτρεμισμό, γιατί ριζοσπαστική είμαι και εγώ και όσο θυμώνω γίνομαι ακόμα πιο ριζοσπαστική. Οπότε καταλαβαίνετε, ακραία πάντως όχι. Πολύ, πολύ μεγάλο δίκιο έχεις λέει ο κύριος Δεπρέ που κάθεται δίπλα της. Ε, έλεγα λοιπόν ε, να σας πω ότι λέει η κυρία Πακάσα Ορτουντούα έχει κάνει τροπολογίες που προσπαθούν να περιορίσουν ε, το εύρος της έκθεσης και το πεδίο εφαρμογής σε σχέση με την αρχική ε, πρόταση. Δηλαδή, ε, επικεντρώνεται πολύ σε κατασταλτικά μέτρα, ενώ η δική μας και ο θέλει να εστιάσει περισσότερο στην πρόληψη. Υπάρχουν και άλλες τροπολογίε για να μην στιγματίζονται ειδικέ κοινότητες με βάση τη θρησκεία τους ή όλες οι δράσεις που πρέπει να αναλυφθούν για να γίνονται πλήρως σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα σχετικά πρότυπα. Η κυρία Παγάσα Ορτοντούα τονίζει επίση τη σημασία τη κοινωνία των πολιτών, όχι μόνο στι τοπικέ κοινότητε, από όπου αρχίζει η στρατολόγηση, αλλά και σε ε, άλλα περιβάλλοντα που αναφέρει, έκθεση όπως είναι σοφρονιστικά καταστήματα, το διαδίκτυο, μήκυο, ε, μπορούν να βοηθήσουν ε, θελοντές, οργανώσει θυμάτων και αστυνομικοί. Επίσης υποστηρίζει ότι η διαδικασία και υπογραμμίζει ότι η διαδικασία στρατολόγησης μπορεί να είναι παγκόσμιο φαινόμενο, δεν θα πρέπει να στιγματίζουμε συγκεκριμένες περιφέρειες ή χώρες, να δούμε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο, αλλά και εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ειδικά σημεία τώρα συγκεκριμένα φυλακές, θέλει να τονίσει τη σημασία των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των σοφρονιστικών υπαλλήλων είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πρακτική άσκηση και εκπαίδευση, όχι μόνο για να ανοιχνεύει κανείς, αλλά και να προλαμβάνει ε, τη ριζοσπαστικοποίηση και μπορεί να είναι καμιά φορά την παραγωγική υπερβολική παρουσία και δίδυση των δημοσίων αρχών. Θα πρέπει να υπάρχει ε, σεβασμός της ελευθερίας της σκέψης και των θρησκευτικών λειτουργών στις φυλακές θέλει να στείλει ένα μήνυμα θετικό για το διαδίκτυο, για τις εταιρείες παρόχους περιεχομένου και τους διαχειριστές. Βεβαίως, αν αρνηθούν τη συνεργασία οι πάροχοι, θα πρέπει να δρούμε, αλλά δεν μπορούμε να θυσιάσουμε την ελευθερία της έκφρασης στο βωμό όλων αυτών. Για την εκπαίδευση, κατά την άποψη της κυρίας Παγάσα Ορτουντούα, αυτό είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο της έκθεσης και ε, αυτό θα πρέπει να τονίσουμε περισσότερο, διότι η ένταξη αρχίζει από εκεί. Δημιουργείται μια θετική αντίληψη για τις κοινέ αρχές και διδάσκουμε ότι οι διαφορές μας μας κάνουν πιο δυνατούς και ε, η ιδέα και η προώθηση της ιδέας της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας είναι ε, κομβικό και κρίσιμο σημείο ειδικά προγράμματα που να εστιάζουν σε θετικές ταυτότητες είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά και πάλι να μην πολύ ανακατεύονται υπερβολικά οι δημόσιες αρχές, είναι σημαντικό αυτό. Και θα πρέπει να εξασφαλίζεται και ελευθερία στην εκπαίδευση και την παιδεία. Και εκπαίδευση, ξέρετε, δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τα σχολεία, αλλά και τις κοινωνίες, τις κοινότητες και τις οικογένειες. Θα πρέπει εκεί από κοινού με εμπειρογνώμονες και οργανώσεις που αφοσιώνονται σε αυτή την προσπάθεια να συνεργαζόμαστε. Και ένα σχόλιο προσωπικό. Έχει μεγάλη ίδια πείρα η κυρία Παγκάσα Ορτούντου με αυτή τη διαδικασία από τη χώρα των Βάσκων. Ένα τελευταίο τονίζει την ανάγκη για ανταλλαγή πληροφοριών και των πρακτικών, καθώς επίσης να πούμε ότι τα ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να γίνονται πάντοτε σεβαστά σε οποιαδήποτε ε, τέτοια περίπτωση που αφορά πολίτες, η στρατολόγησή τους πρέπει να γίνονται πάντα σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ Σοφή. Και τώρα κανονικά το λόγο έχει η συνάδελφος Πινέλη. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την κυρία Γασινταντατή για την ε, πολύ καλή και δύσκολη εργασία που χρειάστηκε να κάνει. Θα μιλήσω ιταλικά όμως τώρα, γιατί και εγώ έχω γράψει κάποιες σημειώσεις εδώ πέρα στα ιταλικά. Ως ασκιώδης λοιπόν η συγγήτρια για τη δική μου την πολιτική ομάδα, ζήτησα μια γνωμοδότηση από 14 μη κυβερνητικέ οργανώσει, τι οποίε και έλαβα, και ουσιαστικά εκφράζουν τι ίδιε πάνω κάτω ανησυχίε για τρία σημαντικά ζητήματα. Η έκθεση, και αυτό λένε οι μη κυβερνητικέ οργανώσει, επικεντρώνεται κυρίω σε μέτρα καταστολή και όχι τόσο σε μέτρα πρόληψη. Και γίνονται πολλές επιθέσεις όχι μόνο από ξένους μαχητές, αλλά στην καρδιά, στο πλαίσιο των δικών μας κοινωνιών και πολλές φορές ε, γύρω από τις αστικές περιοχές. Και έπειτα γίνεται και μια αναφορά στον θρησκευτικό ρίζοσπαστη, στη θρησκευτική ριζοσπαστικοποίηση και αναφέρονται επίσης και σε επιπτώσεις που αυτό μπορεί να έχει για ενδεχόμενο θρησκευτικό στιγματισμό, ότι ελοχεύει δηλαδή και αυτός ο κίνδυνος. Πρόσφατα είχαμε δύο εκθέσεις της Europol όσον αφορά κάποιες ε, βίες τρομοκρατικές επιθέσεις το 2013-2014. Το 2013 ο εξτρεμισμός, ο θρησκευτικός, η, η παστικοποίησης εμφανίζεται ξεκάθαρα σε δύο επιθέσεις δύο από, σε σύνολο 100 περίπου, ενώ το 2014 οι περισσότερες επιθέσεις δεν είχαν θρησκευτικό χαρακτήρα. Αυτό το λέει το ίδιο η Ευρωπόλ. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα προτιμούσα ακόμα και από γλωσσικής πλευράς και συμφωνώ μετά όσο είπε η κυρία Ινβέλτ πριν από μένα, θα προτιμούσα λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε πιο συγκεκριμένους όρους Ακόμα και αν φαίνονται κάπως γενικοί, πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Καλύτερα βίαιος εξτρεμισμός από το να λέμε ρίζος παστικοποίηση ή βίαιος φονταμενταλισμός. Ξέρετε ότι ένας φονταμενταλιστής μπορεί να μην είναι καν βίος. Επομένως δεν θα πρέπει να το στιγματίζουμε. Έχω επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα σημεία στις τροπολογίες μου Αναφέρομαι στην κεντοποίηση και στον κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς επίσης και στην περιθυροποίηση ορισμένων ατόμων, οι οποίοι αισθάνονται όλο και περισσότερο απομονωμένοι από την κοινωνία, ενώ αντίθετα θα πρέπει ουσιαστικά να τους βοηθούμε να ενταχθούν περισσότερο. Επίσης αναφέρομαι και εγώ στο διαχωρισμό που προτείνεται για τα σοφρονιστικά ιδρύματα. Ήδη στα πλαίσια της Επιτροπής μας το είχαμε θίξει το ζήτημα αυτό και τότε η κυρία Ντατή μας είχε πει ότι αυτή αντιμετωπίζει με έναν τρόπο λίγο πιο πολύπλοκο το ζήτημα του διαχωρισμού. Παρ' όλα αυτά σε όλες τις γλωσσικές εκδοχές βλέπουμε τη λέξη, τον όρο διαχωρισμός ή απομόνωση. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να βρούμε έναν άλλον όρο, αντικείμενο συμβιβασμού ενδεχομένω. Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε και εδώ τους σωστούς όρους. Όσον αφορά τώρα το διαδίκτυο, και το ζήτημα αυτό είναι πολύ ευαίσθητο για τη δική μας την πολιτική ομάδα. Οποιαδήποτε λογοκρισία ή οποιοδήποτε έλεγχος θα πρέπει πραγματικά να αποτελεί αντικείμενο πολύ προσεκτικής εξέτασης. Θα πρέπει να εφίστανται όλα τα εχέγγυα για την ελεύθερη έκφραση και το δικαίωμα της επικοινωνίας. Επίσης, Λέμε επίσης ότι θα πρέπει να προωθούμε περισσότερο τη διαφορετικότητα, την ανεκτικότητα και κάτι το οποίο με αφορά ιδιαίτερα. Η δικαστική συνεργασία με τρίτες χώρες. Ζητάω λοιπόν σε μια τροπολογία μου οποιαδήποτε συμφωνία που έχουμε με τρίτες χώρες να περιλαμβάνει συγκεκριμένα ευρωπαϊκά πρότυπα ή και διεθνή πρότυπα πολλές φορές υψηλότερα από αυτά τα οποία προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να υπάρξει οποιαδήποτε σύγχυση μεταξύ τρομοκρατίας και μετανάστευσης και δεν νομίζω θα πρέπει να υπάρξει σε καμία περίπτωση φιλετικό ή εθνικό προφάιλινγκ. Πιστεύω και εγώ ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε έναν κάποιον συμβιβασμό, τουλάχιστον σχετικά αφορά τους όρους που χρησιμοποιούμε, και ελπίζω να ληφθούν υπόψη οι περισσότερες τροπολογίες που έχει υποβάλει η ομάδα μου. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ κυρία Σφινέλη. Η Τζιν Λάμπερτ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Ντατή για την έκθεσή της. Ε, πιστεύω ότι θα μας ε, απασχολήσει αρκετά το καλοκαίρι. Ε, η έκθεση θα μας πάρει χρόνο να δούμε όλες αυτές τις τροπολογίες. Έχουμε ένα ευρυφάσμα επιλογών. Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι το ζήτημα μπορεί να λυθεί εντελώς εντός εθνικών συνόρων με μέτρα καταστολής, ενώ άλλοι έχουν θετήσει μια πιο ολιστική προσέγγιση. Και προείπαν συνάδελφοι ότι θα πρέπει να γίνουν επιλογές. Ήδη βλέπω από τις τροπολογίες ποια είναι αυτά τα σημεία Κάποιες μάλιστα τροπολογίες είναι καλύτερες και από τις δικές μου. Σίγουρα μπορούμε πιστεύω να καταλήξουμε σε συμφωνία μεταξύ μας. Σε σχέση με ορισμένα από τα σημεία που ήδη έχουν τεθεί, πιστεύω και εγώ ότι πρέπει να υπάρξει ε, σαφήνεια για το θέμα. Τι, γιατί μιλάμε εδώ. Έχω καταθέσει και άλλα από την ομάδα μου, όπως τροπολογία 21, για το τι θεωρούμε ότι θα πει ρίζος παστικοποίηση σε αυτό το πλαίσιο για το θέμα των αλλοδαπών ε, μαχητών. Ξεχνάμε ότι πρόκειται συχνά για επικός χωρών της Ένωσης, που επιτίθενται σε άλλους επικούς χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, το πεδίο εφαρμογή γνωρίζω ότι ίδια η έκθεση φιλοδοξεί να έχει ένα ευρύ πεδίο. Εγώ έχω καταθέσει κάποιες τροπολογίες, έχω παραδείγματο χάρη την 142 και την 23. Θέλω να διευκρινίσω τι συζητούμε εδώ υπό την έννοια της ρίζοσπαστικοποίηση. Δεν μιλάμε για μία πίστη ή μία ιδεολογία μόνο υπήρξαν ρατσιστικές επιθέσεις και κατά μουσουλμάνων, ε, είχαμε ισλαμοφοβικές, αντισημιτικές επιθέσεις και άλλες. Είδαμε και ε, φρικαλαιότητες ε, στον υπόγειο του Λονδίνου και τα λοιπά. Είναι λοιπόν αυτές οι επιθέσεις από τελείως διαφορετικά μεταξύ τους άτομα, τελείως διαφορετικά υπόβαθρα, πιστή και επιθήσεις. Επομένως πρέπει να είναι ξεκάθαρο αυτό. Πρέπει να το έχουμε κατά νου, διότι σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να αφήσουμε ορισμένους ε, ελεύθερους και άνετους να οργανωθούν. Επίσης, έχουμε αυτούς που είναι υπεύθυνοι για την ε, παρακολούθηση αφενός και αυτούς ε, που είναι υπεύθυνοι για τη στήριξη αφετέρου. Υπάρχουν κάποιες διακρίσεις και κάποιες γραμμές διαχωριστικές αν βάλουμε κάποια άτομα στο κύκλωμα τη παρακολούθησης περισσότερο, χάνεται η αξιοπιστία, πιστεύω, και αποδυναμώνεται και ο κοινωνικό συστός. Δεν πρέπει να κάνουμε αυτή τη διάκριση πάρα πολύ σαφή τώρα. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι ε, στηρίζουν ε, τον, ε, την τρομοκρατία. Δεν είναι το ίδιο με αυτούς που προσπαθούν να εξηγήσουν τι είναι τρομοκρατία. Αυτό γίνεται στις, ε, αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή έχουμε ένα διάλογο για το τι ε, είδους αφήγηση είναι αποδεκτή στα πανεπιστήμια, ε, μεταξύ των ακαδημαϊκών κτλ. Και τι δεν είναι. Ώστε να μπορούμε να αντικρούσουμε εξτρεμιστική, την εξτρεμιστική αφήγηση, αλλά να προστατεύσουμε ταυτόχρονα και τις θεμελιώδεις οικουμενικές αξίες. Έχω καταθέσει και για τα σοφρονιστικά ιδρύματα τροπολογίες. Θα επανέλθουμε, θα τα συζητήσουμε και ε, στο πλαίσιο της προσπάθειας αναζήτησης συμβιβασμού για το διαδίκτυο επίσης. Σημείο αναφορά για εμά είναι η φυστάμενη νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε τα παιδικής πορνογραφία. Πρέπει να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο. Όχι ανεπίσημα άτυπα να βρουν κάποιες οργανώσεις ώστε να υπάρξει δυνατότητα νομικής προσβολής ή κατάχρησης. Σε ό,τι δεν αφορά τη συνεργασία με τρίτες χώρες, πιστεύω ότι θα πρέπει και εδώ να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή στις ασφαλιστικές δικλίδες. Με τον Κουαντάναμο και άλλα μάθαμε ότι τελικά κατάλαβαν και οι Αμερικανοί ότι ήταν ένας τόπος στρατολόγησης τελικά τον Κουαντάναμο. Και πρέπει να το έχουμε και αυτό υπόψη μα στο πλαίσιο τη συνεργασία με τρίτε χώρε, όπω επίση το ζήτημα τη επιστροφή και επανένταξη. Πρέπει να δούμε τι διδάγματα αντλούν και να μην μείνουμε σε κάποιε προκαταλήψει όπω μπορεί να βλέπουμε με κάποιε τροπολογίε. Πολύ καλή δουλειά έχει γίνει και θα πρέπει να γίνει και βέβαια δεν ζηλεύω καθόλου την εισηγήτρια που θα πρέπει να προσπαθήσει να βρει συμβιβασμού με όλες αυτές τις τροπολογίες που πραγματικά είναι πάρα πολύ πλούσιες. Σίγουρα πάντως θα εργαστούμε επικοδομητικά για να έχουμε την τελική έξι. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, συνάδελφος. Ε, ε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να πω ότι η έκθεση είναι η σημαντικότερη έκθεση που διάβασα το τελευταίο διάστημα. Συνοψίζοντας πρέπει να σας πω ότι καταβάλλεται εδώ μια απόπειρα να εξασφαλιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπήρξαν κάποιοι συνάδελφοι που ανέφεραν ότι ε, έχει αυξηθεί ο αριθμός των ξένων ε, μαχητών. αυτό είναι λόγω των πολλών πολέμων και των πολλών τρομοκρατικών οργανώσεων. Σας δείχνω εδώ μια φωτογραφία, είναι δύσκολο να τη δούμε. Ε, αυτοί είναι οι μαχητές. Ε, είναι πέντε άντρες εδώ, δεν ξέρω αν βλέπετε μακριά τη φωτογραφία. Τρομοκράτες, οι οποίοι Ε, προσπάθησαν και μπορείτε να το δείτε και στο διαδίκτυο. Είναι ένα βίντεο κλιπ που μπορείτε να το δείτε το φιλμάκι αυτό ε, στο διαδίκτυο που έκαναν μια απόπειρα και πραγματικά εγώ όταν το είδα με πιάσαν τα κλάματα. Και ε, βλέπουμε τι γίνεται με τα μεταναστευτικά κύματα που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με διάφορες ε, ανταλλαγές ε, απόψεων ε, που είχαμε καταλάβαμε ότι υπάρχουν προβλήματα και από τις απόπειρες και τις επιθέσεις στο Ρονδίνο, στην Τινησία, στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι βλέπουμε ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα σε μετανάστευση και τρομοκρατία. Πόσοι τρομοκράτε θα πρέπει να φτάσουν ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσα τρομοκρατικά χτυπήματα μέχρι να μπορούν οι πολίτες να ζουν ελεύθερα και ασφαλώς. Ευχαριστώ, συνάδελφο Πάτρου. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση αναφέρεται στην ρίζοσπαστικοποίηση, σαν να ήταν ένα φθόρμητο φαινόμενο, χωρίς κανένα λόγο, χωρίς αιτία. Μα όλοι οι τρομοκράτε χρειάζονται μια κάποια ιδεολογία, μόνο και μόνο ενδεχομένω για να δικαιολογήσουν τις βίες πράξεις τους. Αυτό έχουμε δει τον τελευταίο αιώνα με τους Βάσκους, τους Ιρλανδούς και τις βιοπραγίες που έχουν κάνει πολλές φορές πολλές φορές έχουν προσπαθήσει να δικαιολογήσουν την ε, βίαιη αυτή στάση τους βασιζόμενοι σε συγκεκριμένους πολιτικούς στόχους. Αυτό γίνεται και συγκεκριμένη περίπτωση. Βλέπετε ότι το Ισλαμικό κράτος θέλει να δημιουργήσει ένα χαλιφάτο και ότι θα θέλουν να επιβάλλουν τη θρησκεία τους παγκοσμίω. Έτσι δικαιολογούν την τρομοκρατική τους ε, δράση. Στην έκθεση αυτή δεν αναφέρεται ούτε το Ισλάμ, ούτε οι τζιχαντιστές, αναφέρονται ευτυχώς στις τροπολογίες που έχουμε καταθέσει. Όλοι αυτοί οι τρομοκράτες έχουν το εξής κοινό. Διαβάζουν όλοι το ίδιο βιβλίο, το Κοράνι, το οποίο σε κάποια σημεία λέει σκοτώστε τους άπιστους όπου τους βρείτε, ε, προσπαθήστε να τους τρομοκρατήσετε, κάντε τρομοκρατικές επιθέσεις στις χώρες τους κτλ και λέγεται επίσης ότι η μέρα της κρίσης δεν θα έρθει παρά μόνο την ημέρα που οι α, μουσουλμάνοι θα καταφέρουν να νικήσουν, να κάνουν πόλεμο εναντίον των Εβραίων. Επομένως, όντως, μιλάμε αυτή τη στιγμή για δύο εξτρεμισμό και μιλάμε για μια στρατιωτική εκδοχή, αν θέλετε, του μουσουλμανισμού και είναι, αν θέλετε, το πιο ακραίο παράδειγμα το οποίο έχουμε όταν άνθρωποι σκοτώνουν, αυτοκτονώντας οι ίδιοι, γιατί θα πάνε στο παράδεισο όπου τους περιμένουν πάρα πολλές παρθένες. Επομένω, πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε καταρχάς την ιδεολογία που διέπει όλες αυτές τις πράξεις. Και υπάρχει εδώ πέρα μία αντιπαράθεση ανάμεσα στους μετριοπαθείς και τους πιο ακραίους. Ο βασιλιάς της Ορδανίας που ήρθε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας είπε ότι ακριβώς υπάρχει μία μάχη, πρέπει να διεξαχθεί μία μάχη ανάμεσα στους μετροπαθείς και τους ακραίους. Και οι μετροπαθείς θα πρέπει να καταφέρουν να, να παραμερίσουν στο Κοράνι όλους, όλες αυτές τις ακραίες δηλώσεις που γίνονται και θα πρέπει να καταφέρουν να διώξουν από τα τζαμιά τα πιο ακραία στοιχεία. Και οι δυτικέ κυβερνήσει από την άλλη θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν ότι το φονταμε, ο φονταμεταλισμός στα πλαίσια του Ισλάμ δεν έχει καμία θέση στις δυτικές κοινωνίες. Στην πράξη όμω τι μπορούμε να κάνουμε για να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Νομίζω θα πρέπει να σταματήσει καταρχά η μαζική μετανάστευση. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να την επιταχύνουμε όπω είπαμε σήμερα το πρωί και να βρούμε νέου νόμιμου τρόπου για να προσελκύσουμε περισσότερου μετανάστε. Δεν καταφέρνουμε καν να ενσωματώσουμε όλου αυτού που ήδη βρίσκονται στι χώρε μα και δεν εστερνίζονται την δυτική αντίληψη και το δυτικό πολιτισμό. Θα πρέπει να σταματήσουμε επίση τη χρηματοδότηση τζαμιών και ημάμιδων από το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία, οι χώρες που δίνουν πάρα πολλά χρήματα προκειμένου να οικοδομηθούν τζαμιά, τζαμιά και να διοριστούν νέοι μάμιδε. Αυτό βλέπω και στο Ανατολικό Λονδίνο, τη δική μου την εκλογική περιφέρεια. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Και πρέπει επίση να αλλάξει η κοινοτροπία, η όλη αντίληψη που έχουν οι άνθρωποι αυτοί. Αλλά πρώτα πρέπει να αλλάξει η δική μα η αντίληψη. Θα πρέπει εμεί ε, ω Δύση να σταματήσουμε να ευνοούμε ουσιαστικά αυτή την ανοτροπία του Μεσαίου να τρέφουν ορισμένοι άνθρωποι. Ευχαριστώ, συνάδελφος Μάγια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι ε, πραγματικά πάρα πολύ επίκαιρη έκθεση. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες. Ε, είναι πολύ δύσκολο ε, να μιλάς για μια τέτοια έκθεση χωρίς να λες τα πράγματα με το όνομά τους. Ο Ισλαμικός ε, ε τρόπος ε, τρομοκρατίας, Ισλαμική τρομοκρατία βρίσκει πρόσφορο έδαφος ε, νέους που δεν αισθάνονται καλά, δεν είναι καλά στη ζωή τους και υπάρχει ιδεολογία από πίσω που λέγεται το Ισλάμ. Θέλω να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, να μην ε, χρησιμοποιούμε περιστροφές και να μην αποφεύγουμε την ουσία. Δεν πρόκειται να είναι πιο ασφαλής ο κόσμος. Ε, αντί να προλαμβάνουμε ε, την επιστροφή των τρομοκρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εστιάζεται στο να μην τους αφήνουμε να φεύγουν. Εγώ προτιμώ να φύγουν παρά να παραμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 5.000 λέει τζιχαντιστές έχουν φύγει στο μεταξύ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσοι γύρισαν, άλλοι τόσοι και πού βρίσκονται αυτοί. Έχουμε καμιά ιδέα, ε, τους έχουμε εντοπίσει και βλέπω και στην έκθεση να μιλάτε για έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα. Αλλά όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, φέρνει καραβιές ε, με παράνομους μετανάστες, που ε, ξέρουμε αν υπάρχουν μέσα Ισλαμιστές, τι κάνουμε, μια τρύπα στο νερό. Θα πρέπει να ξεφύγετε αυτά που λέτε ε, για τους ημάμιδες ε, ε, που διαδίδουν και κάνουν κηρύγματα μίσους. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους τσιχατιστές που επιστρέφουν και να κλείσουμε τα σύνορα με ριζικά μέτρα και να επανέλθουν οι έλεγχοι στα σύνορα, όπως κάνει η Αυστραλία που τους στέλνει από εκεί που ήρθανε. Ένας τελευταίο συνάδελφο ακόμα στη λίστα των ομιλητών είναι ο συνάδελφο Ζεγάρ Δεπχέ. το λόγο Ζεγάρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι αρκετά σύντομο. Καταρχά, θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Ντατή για την έκθεσή τη, παρόλο που έχουμε κάποιοι από εμά επιφυλάξει και είναι φυσιολογικό αυτό για τι προτάσει ορισμένοι θέλουν να βάλουν κάποιες αποχρώσεις. Πάντως η έκθεση είναι πολύ καλή ως βάση εργασίας γιατί σαρώνει ε, όλο το πεδίο και θέτει ε, τις σωστές βάσεις. Και θα ήθελα να σας πω κύριε Συγκήτρια, μην αφήνετε να σας ε, παρενοχλούν ή να σας αποσπούν εκείνοι που σας κατηγορούν για ε, συμπάθεια των ε, τρομοκρατών. Είναι μάλλον η λυθιότητα αυτό παρά σοφία και μετράω τα λόγια μου. Και γίνονται και συγχύσεις μεταξύ των παράτυπων μεταναστών. Μπορεί να υπάρχουν τρομοκράτες, αλλά δεν είναι όλοι τρομοκράτες. Προσοχή λοιπόν να μην πέφτουμε σε τέτοιες απλουστεύσεις και σε απλή βλακεία, εν πάση περιπτώσει. Ε, έχουμε κάνει τροπολογίες ε, που έχουν τέσσερις στόχους, κυρία Συγήτρια. Μιλάτε πάρα πολύ για στρατηγική. Αυτό δικεί λίγο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί επανειλημμένα ε, έχει ορίσει η Στρατηγική Επιτροπή και μάλιστα την ενημερώνει αυτή τη στρατηγική. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο δράσης. Η στρατηγική είναι δεδομένη, η υλοποίηση είναι τώρα, η εκτέλεση το θέμα του εκτελεστικού επιχειρησιακού σχεδίου, γιατί έχουμε πραγματικές απειλές. Και αυτό θα πρέπει να συγκεντρώσει τη δική μας προσοχή τώρα. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την ορολογία και τις σχετικές συζητήσεις, και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να αναφερθούμε στο σημειωματικό πρωτόκολλο, λέει, του Συμβουλίου της Ευρώπης για δύο εξτρεμισμό και ριζοσπαστικοποίηση που οδηγούν στην τρομοκρατία. Περί αυτού ακριβώς πρόκειται. Ε, και τρίτον, είμαι μεταξύ εκείνων που θέλουμε να ενισχύσουμε το ρόλο της Ευρωπόλ. Ιδιαίτερα για την καταπολέμηση του επικινδύνου και τρομοκρατικού περιεχομένου που ανθεί στο, κοινοβούλιο, στο διαδίκτυο. Συγγνώμη. Ε, ακούω πολλά για τα τζαμιά αλλά ε, το διαδίκτυο επηρεάζει περισσότερο τους νέους. Το ίντερνετ τα μαθαίνουν αυτά, όχι στο τζαμί. Και εκείνοι που πάνε στο τζιχάτ στη Μέση Ανατολή έχουν επηρεαστεί περισσότερο από τα tweets, τα τετιβίσματα των φίλων τους, από το ίντερνετ και λιγότερο από το τέμενος που δεν πατάνε κιόλας. Ε, το θέμα μπορεί να είναι ε, λεπτό και ευαίσθητο, το ξέρω, γιατί είναι λεπτή η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα ε, στην ελευθερία της έκφρασης και στην υποδάβηση του μίσου ή στην υποκίνηση για δολοφονίες. Αν έχω σωστές πληροφορίες από την αρχή του μηνός Ιουλίου, υπήρξαν 50 επεμβάσεις σε site, ε, στο Twitter ή αλλού που ε, έχουν απαλληφθεί χάρη στην παρέμβαση της Ευρωπόλ που είναι πιο αποτελεσματική εδώ από το άθροισμα των κρατών μελών. Ξέρω ότι είναι το θέμα λεπτό αυτό και ευαίσθητο, ήθελα να το πω. Τέταρτο και τελευταίο, Συμφωνώ με κάποιους προλύσαντε συναδέλφου, Δεν θα πρέπει απλώ να εκφράζουμε την ανησυχία μα για το τι συμβαίνει στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει και εξωτερική στρατηγική που έχει μεγάλη σημασία και πρέπει να βοηθήσουμε κάποιε από τι χώρε εταίρου που είναι ιδιαίτερα τώρα ευάλωτε να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να καταπολεμήσουν την ριζοσπαστικοποίηση της δικής τους νεολαίας. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή να χορηγήσει περισσότερα κονδύλια στη βοήθεια των χωρών αυτών για να ε, πάνω στα χέρια τους το μέλλον των νέων τους και να καταπολεμήσουν ε, την ε, υποκίνηση του μίσους για τη βία και για το τζιχάτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δώσετε το λόγο. Εγώ ευχαριστώ Ζεράρ. Πολύ σύντομα η συνάδελφος Κιένγκε τελευταία και μετά η κυρία Ρασιντά. Τότε εισηγητή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το ζήτημα που συζητάμε είναι πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον. Εγώ ασχολούμαι με το ζήτημα αυτό στην Επιτροπή Πολιτισμού και συμμετέχοντας και στην Επιτροπή αυτή, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να δούμε πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε ακόμα και την πολιτική διάσταση στο ζήτημα αυτό. Είναι πολύ σημαντικός ο πολιτισμός για την απορίζοσπαστικοποίηση. Δεν θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε μόνο σε αρνητικές πτυχές, αλλά και στην πιο θετική εξέλιξη. Πώς μπορούμε να οδηγηθούμε δηλαδή σε μια απορίζοσπαστικοποίηση που να εμπλέκει βέβαια και τους ενδιαφερομένους, αλλά και τις οικογένειές τους. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε να στηρίξουμε τις ίδιες τις οικογένειες των ανθρώπων αυτών, πώς μπορούν να συμβάλλουν ώστε να απορροσπαστικοποιηθούν προκειμένου να αποφύγουν οποιοδήποτε φαύλο κύκλο. Πέρα όμως από τις οικογένειες πρέπει να υπάρχει και ένα ολόκληρο δίκτυο για να υποστηρίξει και να βοηθήσει τα άτομα αυτά, κυρίως ένα δίκτυο μέσω από το σύστημα παιδείας, μέσω των σχολείων, μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων εκπαιδευτικών, αλλά και μέσω πολιτισμικών προγραμμάτων στα σοφρονιστικά ιδρύματα. Εκεί δηλαδή όπου όντως έχουμε πολλά υψηλά ποσοστά ρίζοσπαστικοποίησης. Πρέπει να έχουμε λοιπόν κάποια κατά περίπτωση ad hoc προγράμματα, τα οποία να έχουν τόσο πολιτισμική όσο και ψυχολογική διάσταση, προκειμένου να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι πολύ συχνά οι οποίοι όταν θα βγαίνουν από αυτά τα προγράμματα από οροσπαστικοποίησης να μπορούν και οι ίδιοι με τη σειρά τους να βοηθήσουν άλλους ρεσπαστικοποιημένου νέους για να βγουν από αυτό το φαύλο κύκλο. Και κάτι το οποίο παρατήρησα Αναφερόμαστε πολύ στο πώς θα καταφέρουμε να ταυτοποιήσουμε και να αναγνωρίσουμε τα άτομα αυτά. Αλλά ας μην υπεργενικεύουμε, γιατί πολλές φορές αυτό ακριβώς γίνεται. Δημιουργούμε κάποια στερεότυπα για τους ανθρώπους αυτούς και πολλές φορές θεωρούμε ότι βρίσκονται στα, στους κύκλους των μεταναστών ή των λιγότερο προνομίουχων ανθρώπων. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί κάθε φορά που κάνουμε κάτι τέτοιο. Ας μην υπεραπλουστεύουμε, δεν είναι οι άνθρωποι αυτοί αναγκαστικά άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στις πιο φτωχές, στις λιγότερο προνομιούχες κοινωνικές τάξεις. Ξέρετε ότι πολλές φορές υπάρχουν ρεσπαστικοποιημένα άτομα τα οποία δεν προέρχονται από μειονεκτούσες κοινωνικές τάξεις, αλλά που έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από αυτά που διαβάζουν στο διαδίκτυο. Ας μην έχουμε λοιπόν προκαταλήψεις ως προς αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι η συζήτηση που γίνεται εδώ πέρα στη ΛΥΜΠΕ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την πολιτισμική και την εκπαιδευτική διάσταση της αντιμετώπισης του ζητήματος. Και κατά αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε έμφαση τα συστήματα παιδείας, τα οποία θα πρέπει να είναι περισσότερο διαπολιτισμικά. Να καταφέρουμε δηλαδή μέσω της προσέγγισης αυτής και μέσω της ε, γνώσης των άλλων πολιτισμών και των άλλων θρησκειών, να καταφέρουμε να απομακρύνουμε όλα αυτά τα φαινόμενα φόβου και να καταφέρουμε κατά αυτόν τον τρόπο να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Μόνικα να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους. Θα είμαι πιο σύντομη γιατί συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Και με την ορολογία, του ορισμού συμφωνώ με τους κύριες Γκόμες, ε, Σπινέλη, Ιντβελ, τον κύριο Ντεπρέ. Πράγματι ε, πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Πράγματι υπάρχει ριζοσπαστικοποίηση ε, ή φονταμενταλισμός ισλαμικός. Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι μπορούμε να το ταυτίσουμε με τους τρομοκράτες ή τους διχατιστές και όσο πιο ασαφείς είμαστε τόσο λιγότερο θα είμαστε αποτελεσματικοί για τη στρατηγική θα πρέπει να υιοθετήσουμε ένα συνεκτικό πρόγραμμα δράσης ε, πρέπει να μετατοπίσουμε το βάρος μας ε, από τη στρατηγική στο πρόγραμμα δράσης για τους κρατουμένους. Πράγματι, ε, ούτε θέλω την ε, απομόνωση, ούτε το διαχωρισμό για τους κρατουμένους αυτούς. Ε, απλά στη Γαλλία γίνεται ένα πείραμα, είναι πολύ αποτελεσματικό και μάλιστα επανεντάσσονται κάποιοι από τους κρατούμενους που απλά είναι κάπως ευαίσθητοι και θέλουν να ριζοσπαστικοποιηθούν, αλλά τελικά δεν είναι αυτό το πρόβλημά τους. Ε, και πράγματι συμφωνώ ότι πολλά γίνονται στο διαδίκτυο και πολύ λιγότερα στα τεμένη. Πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία. Ναι, καταλαβαίνω και τα περί έκφρασης και λοιπά. Όμως πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί απέναντι στο διαδίκτυο ε, από αυτούς που εποφελούνται και για να κερδίσουν χρήματα από το μέσο αυτό. Τώρα, καταστόλη, ναι, χρειάζεται ε, τα προτινόμενα μέτρα είναι σημαντικά, αλλά και η πρόληψη είναι εξίσου σημαντική. Η έκθεση θα πρέπει πράγματι να περιλαμβάνει και αποτελεσματικά προληπτικά μέτρα για το ρόλο της Ευρωπόλου. πολύ σημαντικός, είναι ένα καλό εργαλείο, ένα καλός ε, ε, μηχανισμός, ε, το όργανο αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά και την τρομοκρατία και τη ριζοσπαστικοποίηση. Εξωτερική χρηματοδότηση, ε, το είχαμε πει μάλλον με την κυρία Γκόμες την τελευταία φορά, πρέπει να δώσουμε περισσότερο έλεγχο, περισσότερη χνηλασιμότητα για τις εξωτερικές συναλλαγές και να δούμε ότι κάποιες χώρες όπως η Ειδική Αραβία παίζουν διπλό παιχνίδι. Πράγματι ισχύει αυτό και ε, δεν πρέπει να είμαστε υποκριτέ. Γιατί είμαστε υποκριτέ, συνεργαζόμαστε με χώρε σαν αυτήν, αλλά από ε, σε ό,τι έχει να κάνει με τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα όχι. Αλλά μιλάμε για ε, τρομοκρατική, είπατε μετά ε, και εσείς για, για το Λονδίνο. Ναι, πράγματι υπάρχουν ε, τρομοκρατικά κυκλώματα που τρο, τροφοδοτούνται, χρηματοδοτούνται από αυτές τις χώρες. Ε, για τις ε, συμβαστικές νομίζω θα συμφωνήσουμε. Θα ήθελα επίσης να απαντήσω Μίλησε για βλακεία ο κύριος ε, Ντεπρέ. Εγώ θα έλεγα να πάψουν και οι ύβρις και ο στιγματισμός. Ε, έχουμε δει ε, κάποια στερεότυπα που μπορούν να οδηγήσουν. Δεν πράγματι, το να λέμε μετανάστης ο τρομοκράτης, ε, είδαμε που οδήγησε, είμαι πολύ κατά. Υπάρχουν κάποιοι ε, μετανάστες που έχουν κάνει τρομοκρατικές επιθέσεις, ε, αλλά να μην γενικεύουμε. Θα είναι πολύ καλύτερο αυτό και ε, θα είμαστε και πιο αποτελεσματικοί, θα μας ακούσουν περισσότερο αν αποφεύγουμε υπερβολές και γενικεύσεις όπως αυτά που ακούμε εδώ και χρόνια. Τρομοκράτες ότι είναι θύματα. Πού το λέμε αυτό. Φυσικά, σεβασμός θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η βαρβαρότητα δεν μπορεί να αντικρουστεί με βαρβαρότητα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για οδόντα αντιοδόντος. Και για τους ε, κρατούμενους ε, του Γκουαντάναμου, για παράδειγμα. Για κάποιου δεν υπήρχε καμία κατηγορία. Φεύγουν από εκεί, έχουν ριζοπαστικοποιηθεί και κάνουν τρομοκρατικέ επιθέσει. Άρα, μήπω και εμεί πρέπει να δείξουμε περισσότερη υπευθυνότητα. Και εμεί, Ευρωβουλευτέ, είμαστε σε ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο και ξέρουμε ότι το κράτο δικαίου, τα θεμέλια δικαιώματα μα επιτρέπει να μπορέσουμε να συζητούμε δημοκρατικά εδώ. Αυτά είχα να πω. Νομίζω ότι και με τη σημερινή συζήτηση ε, φαίνεται ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς και να έχουμε και ένα σχέδιο δράσης ε, από τώρα μέχρι το Σεπτέμβριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία. Είναι πάνω από 662 οι τροπολογίες και καλή επιτυχία να τα συγκεράσετε όλα αυτά. 12 και 13 Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή μας, ενώ στην Ολομέλη έχει προβλεφθεί για τη δεύτερη, μάλλον για τον Νοέμβριο του 2015. Επόμενο θέμα, 19, ε, έχει αναβληθεί κοινή συνενέση, οπότε πάμε στο 20, ε, ρώτηση με έτοιμα γραπτής απάντηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της 12ης Μαρτίου σχετικά με τα χρήματα που δαπανώνται για τη Frontex στην Ισπανία εκ μέρου της κυρίας Μαρίνα Αλμπιόλ Γκουσμάν. Θα μας την παρουσιάσει αγαπητοί συνάδελφοι. Σύμφωνα με το άρθρο 134 του, κανονισμού, 130 παράγραφος 4 του κανονισμού, ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιος είναι ο κ. Βόιτσοκ Θαλοτσίνσκι. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Good afternoon. Χαίρετε. Η Βόητε καλωσίσκη από τη Γενική Διεύθυνση ε, Μετανάστευσης και Εσωτερικών και διαχείριση Συνόρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να δώσω απάντηση στη γραπτή ερώτηση που υποβλήθηκε για τον προπολογισμό της Frontex. Θα ήθελα να σας εξηγήσω ότι η ερώτηση αυτή αφορά την υλοποίηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού της Frontex και σύμφωνα με την πρακτική που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβιβάσαμε την ερώτηση για λεπτομέρειες. Η απάντηση εστάλει στις 18 Ιουνίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έδωσε η Frontex η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε επιστολή στην αξιότιμη κυρία Βουλευτή μια συμπληρωματική απάντηση με όλα τα στοιχεία. Θα ήθελα να συνοψίσω τα στοιχεία αυτά, ε, όπως ήδη ε, αναγράφονται στην ελόγω επιστολή. Σύμφωνα με τη χρηματοδότηση ε, στις επιχειρήσεις στην Ισπανία της Frontex, θα ήθελα να τονίσω ότι έχει συντονίσει και συγχρηματοδοτήσει τέσσερις κοινέ επιχειρήσεις στην Ισπανία το 2014, Ήρα, Ινταλάο, Μινέρβα και focal point C. Αυτές είναι οι τέσσερις. Τα συνολικά ποσά ε, ήταν 4.681.000 ευρώ. 4.681.000. Σε ό,τι αφορά τη χρήση και τη δαπάνη αυτή και το σύστημα ελέγχου, η Frontex έχει ένα σύστημα υγιές για τον έλεγχο ε, το λογιστικό έτσι ώστε τα χρήματα που δεσμεύονται για συγκεκριμένες επιχειρήσεις να χρησιμοποιούνται με χρηστό τρόπο. Και επειδή ε, το λέει και η γραπτή ερώτηση, το Mos Majorum που ήταν μια επιχείρηση στην οποία αναφέρεται η κυρία Βουλευτής ε, οργανώθηκε και εκτελέστηκε από Ιταλικές αρχές κατά τη διάρκεια της Προεδρίας και δεν συμμετείχε καθόλου η Frontex στη χρηματοδότηση σε ό,τι αφορά ε, την εκ αξιολόγηση των κοινών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 33 εδάφιο 3 του χρηματοδοτικού κανονισμού της Frontex θα αξιολογήσει Frontex τα αποτελέσματα όλων των κοινών επιχειρήσεων και όταν κληρωθεί αυτό σε συνεργασία με το λόγο κράτος μέλος και τα άλλα κράτη-μέλη που συμμετέχουν ε, γίνεται μια τελική έκθεση αξιολόγησης από τη Frontex. Κατά τη διάρκεια αυτή εκτελούνται μελέτες και αξιολογήσεις και για την εκτέλεση του προγράμματος και για τα οικονομικά. Αναφέρονται ε, λοιπόν τα στοιχεία και στις τέσσερις αυτές επιχειρήσεις σύμφωνα με την ερώτηση ε, της κυρίας Αλβιόλ ε, τα αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να μπούμε σε όλες τις λεπτομέρειες και στην περιγραφή των στοιχείων. Είμαι σε θέση να σας διαβάσω τα τέσσερα παραρτήματα που επισυνάπτονται. Ε, όχι βέβαια. Κύριε Ντεπρέ, η κυρία Ελμπιόλ. Εκείνη θέλει, ε, Ζεράρ δεν θέλει. Ε, Ζεράρ την πάτησες. Ωραία. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την Ήρα, 2014 ήταν η κοινή επιχείρηση. Ήταν ε, διάφοροι στόχοι ε, που είχε βασικό στόχος ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων και σύμφωνα με την αξιολόγηση που έκανε ο οργανισμός αυτό επετεύχθη. Επόμενος στόχος ενίσχυση της αποτελεσματικότητας ασφάλειας των συνόρων ε, σύμφωνα με τον οργανισμό αυτό εν μέρη επετεύχθη μόνο. Επόμενος στόχος ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας και αυτό εν μέρη μόνο έχει επιτευχθεί σε ό,τι αφορά την ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών και αυτό εν μέρει επετεύχθη, σε ό,τι αφορά την αυξημένη αποτελεσματικότητα της ανταλλαγής πληροφοριών εντάξει, ενδεχόμενοι κίνδυνοι και απειλές δεν εντοπίστηκαν σύμφωνα με τις πληροφορίες και την ενημέρωση που λήφθη και μας έδωσε η Frontex για την εγκληματική δραστηριότητα και τα δίκτυα που συνδέονται με την παράτυπη μετανάστευση και τις απειλές και τους κινδύνους. Οι τελευταίοι δύο στόχοι είχαν να κάνουν με την ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών. Αυτό εντάξει, επιτεύχθη επίση με τη ε, συγκεκριμένη επιχείρηση και τελευταίος στόχος να υπάρξουν ε, μόνιμες δομές. Και αυτό επιτεύχθη. Σε ό,τι αφορά το Το 2014 άλλη κοινή επιχείρηση. Στόχοι ενίσχυση ασφάλειας σύνορων εντάξει. Στόχος ενίσχυση αποτελεσματικότητας των σύνορων επίσης επιτεύχθη. Άλλος στόχος ενίσχυση επιχειρησιακής συνεργασίας επιτεύχθη. Ε, ενισχυμένη ανταλλαγή προφοριών δεν επιτεύχθη πλήρως αποτελεσματικότητα στην ανταλλαγή προφοριών επετεύθη. Άλλος στόχος να εντοπιστούν κίνδυνοι και απειλές επίσης επετεύθη. Σε ό,τι αφορά τις ε, βέλτιστες πρακτικές, ε, την εγκαθίδρυση και ανταλλαγή τους επίσης, ε, μόνιμες δομές επίσης εντάξει. Και αυτός ο στόχος επετεύχθη. Τρίτη επιχείρηση στην Ισπανία το 2014, επιχείρηση Μινέρβα πρώτος στόχος ε, αύξηση της ασφάλειας των συνόρων. Η αξιολόγηση θεωρεί ότι ε, ήταν ε, τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ασφάλεια των συνόρων και αύξηση της επίσης, στόχος που επετεύχθη. Ενίσχυση επιχειρησιακής συνεργασίας και αυτό ανταλλαγή πληροφοριών. Επίσης θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί ο στόχος ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στην ανταλλαγή ε, των πληροφοριών εν μέρη, ε, εντοπισμός κινδύνων και απειλών, επίσης στόχος που επιτεύχθη, εγκαθίδρυση και ανταλλαγή των πρακτικών και επίσης θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί. Σε ό,τι αφορά την υποστήριξη, την κατάρτιση, εν μέρη επετεύθεως στόχος. Όλα αυτά λοιπόν ήταν τα παραστήματα. Και τελευταία, τέταρτη τώρα επιχείρηση, Focal Point C ήταν κοινή επιχείρηση το 2014, είχε τους εξής στόχους. Άξιση ασφάλειας των συνόρων. Πλήρως είχε επιτευχθεί. Άλλος στόχος, ενίσχυση αποτελεσματικότητας ε, των ε, ελέγχων στα σύνορα εν μέρη ενίσχυση επιχειρηματική συνεργασίας πλήρως, ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών εν μέρη επιτεύχθη σε ό,τι αφορά το στόχο για την αύξηση της ανταλλαγής των πληροφοριών στην αποτελεσματικότητα εν μέρη και ενδεχόμενοι κίνδυνοι και απειλές θεωρήθηκε ότι επίσης εν μέρη επιτεύχθη σε ό,τι αφορά τους στόχους να εγκαθιδρυθούν και να ανταλλάσσονται βέλτιες πρακτικές. επετέφθη πλήρως και ο άλλος στόχος ε, κατάρτιση και εκπαίδευση εν μέρη επετέφθη. Και τέλος θα ήθελα να τονίσω το εξής. Η Frontex είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ιδρυθεί με κανονισμό του Συμβουλίου σύμφωνα με τις ε, πρακτικές ε, τη μόνη ευθύνη για όλα αυτά που σας ανέγνωσα ε, την φέρει αποκλειστικά και μόνο η Frontex. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απλώς διαβιβάζει. Σας ευχαριστώ. Ήταν εξαντλητική για όσο και πληρέστατη η παρουσίασή σας η κυρία Μαρίνα Αλβιόλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για μας η απάντηση είναι τελείως ανεπαρκής όπως καταλαβαίνετε. Το περιμέναμε πρέπει να σας πω, διότι Frontex είναι ένας οργανισμός που λειτουργεί με απόλυτη αδιαφάνεια, σκοταδισμό και δεν επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει τη δουλειά του, να μετράει και ε, τα οικονομικά και τις δαπάνες. Εμείς θέλαμε τα στοιχεία με βάση τους στόχους και με βάση τις συγκεκριμένες δράσεις και όχι αυτά που μας διαβάσατε. Για παράδειγμα, πόσα λεφτά δίνει η Frontex και η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μελίγια, σε αυτό το φράκτη ε, που έχει ξηράφια επάνω και λάμες και σκοτώνει τον κόσμο. Δίνουν εκεί λεφτά ε, ε, που τα χρησιμοποιούν για τις ενθερμό ε, ε, αποθήσεις που παραβιάζει το Σύνταγμα της Ισπανίας, τον ποινικό κώδικα, την οδηγία για τις επιστροφές, για τη μη επαναπροώθηση, για το άσυλο, το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτές οι ενθερμό αποθήσεις παραβιάζουν τη συνθήκη της Γενέβης, το καθεστώς του πρόσφυγα, την οικουμενική διακήρυξη και πάει λέγοντας. Αυτά τα ξέρετε, δίνουμε λεφτά εμείς αυτά στις ενθερμό αποθήσεις που τους πιάνουν πάνω στο φράχτη και τους γυρνάνε πίσω. Yes. Η, η πρόεδρος διακόπτη. Μήπως θα μπορούσατε να μιλάτε λίγο πιο αργά, γιατί και οι διερμηνείς άνθρωποι είναι. Και πραγματικά δεν σας παρακολουθούν με αυτή την ιδιότητα ταχύτητα. Ζητώ συγγνώμη. Έλεγα λοιπόν, γίνονται αυτές οι αποθήσεις εν θερμό, τις οποίες η κυβέρνηση νομιμοποίησε της Ισπανίας, αν μπορεί να νομοθετηθεί ε, τέτοια νομιμοποίηση ενός αθέμητου τρόπου και αυτό απασχολεί τον κόσμο ε, και σήμερα ε, ε, το, Ευρωπαϊκό, το, το Ισπανικό Λαϊκό Κόμμα απέτρεψε τη συζήτηση αυτού του θέματος στην Επιτροπή μας για τον νόμο περί ασφαλείας των πολιτών στην Ισπανία. Γνωρίζετε κι εσείς και εμείς και όλοι ότι δεν ισχύουν αυτά που λέει. Κατάρτιση λέει για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα σώματα ασφαλείας και στις δυνάμεις ασφαλείας. Εμείς πήγαμε στη Μελίγια, κάναμε εκεί συναντήσεις και ε, συσκέψεις και ξέρουμε ότι αυτά δεν συμβαίνουν. Και δεν μπορείτε να μας λέτε ότι είναι στόχος που έχει επιτευχθεί. Αυτό το αποκρούουμε. 4 εκατομμύρια λέτε 681.000 για την προστασία και προάσπιση των συνόρων. Από ποιον κινδυνεύουν τα σύνορα. Είναι εχθρός ο μετανάστης που απειλεί τα σύνορά μας. Και ένα τελευταίο, όλα αυτά τα λεφτά καλά θα κάναμε να τα επενδύουμε ε, σε χώρους και μηχανισμούς για να μπορούν να γίνονται σωστά ε, οι διαδικασίες, η αίτηση για, για διεθνή προστασία, ε, ανθρωπιστική διάδρομη ή να επενδύονται ακόμα σε χώρες προέλευσης και καταγωγής για να αντιμετωπίσουμε τις πολιτικές εκείνες και τις καταστάσεις που καταδικάζουν χιλιάδες ανθρώπους στην προσφυγιά. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ξαναμιλήσει γι' αυτό. Όχι από ό,τι φαίνεται, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν επιθυμεί να επανέλθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε στο επόμενο θέμα, μόνο 21, Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Δομήνικα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχία διαμονή. Η συγκήτρια είναι η κυρία Μαρία Γκαμπριέλ, την οποία δεν βλέπω. Α, καταφτάνει. Εντός των επομένων λεπτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ήδη παρούσα. Μήπως θέλει να μιλήσει πρώτα η Κομισιόν πριν έρθει η συγκήτρια. Irgendwie sind heute Nachmittag auch die Kommission nicht mehr ganz Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι τόσο πρόθυμη. Ποιο είναι αρμόδιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ε, κυρία, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Um, thank you, Madam Chair. ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σα πω ποιο είναι το γενικότερο πλαίσιο για τις προτάσεις αυτές. πρόκειται για συμφωνίες τις οποίες παρουσίασε τον Νοέμβριο του 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πέντε χώρες της Καραϊβικής και 11 νησιά του Ειρηνικού που μπορούν να περάσουν στον ε, κανονισμό αυτό 539 του 2001 που παρέχει την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρηση για βραχία διαμονή. Έγινε λοιπόν μια αξιολόγηση αναπερίπτωση για κάθε χώρα ξεχωριστά, χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένα κριτήρια, ο ενδεχόμενος κίνδυνος παράνομης μετανάστευσης, ε, κάποια κριτήρια που έχουν να κάνουν με τις ε, δημόσιες πολιτικές ασφάλειες, ε, ζητήματα μηδεότητας κτλ. Γίνανε λοιπόν διαπραγματεύσεις με τους συνομοθέτες και σύμφωνα με τον κανονισμό 539 εγκρίθηκε η πρόταση αυτή και έχουμε τις χώρες αυτές από την Καρυβική και τον Ειρηνικό, καθώς επίσης και τα Ενωμένα Αραβικά Μοιράτα, το Περού και την Κολομβία, που δεν είχαν αρχικά προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως χώρες μπορούσαν να περάσουν στο θετικό κατάλογο. Προκειμένου να δοθεί αυτή η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης, από τον κανονισμό που έχει αρχίσει να ισχύει, πρέπει να υπογραφεί μια συμφωνία απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρηση για κάθε μία από τι χώρε αυτέ, προκειμένου να υπάρχει απόλυτη αμοιβαιότητα. Δηλαδή ότι μπορούν και οι πολίτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάνε στι χώρε αυτέ χωρί να απαιτείται και για αυτού για την ίδια χρονική περίοδο θεώρηση. Οι συμφωνίε με νέα χώρε έχουν ήδη υπογραφεί και έχουν προσωρινά τεθεί ενισχύ με τις πέντε χώρες της Καρεβικής, τη Δομίνικα, την Γρανάδα, τη Σάντα Λουσία, το Σαν βινσεντε Τρινιδάτ, το Μπάγκο και επίσης με τη Σαμόα, το Βανουάτου και τον Ανατολικό Τιμόρ και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έχουν ήδη υπογραφεί όλες αυτές οι συμφωνίες με αυτές τις χώρες και έχουν προσωρινά τεθεί ενισχύ και έχουν υποβληθεί συμφωνίες αυτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να δώσει και αυτό την έγκρισή του θα κάνω μια κοινή παρουσίαση για όλες αυτές τις περιπτώσεις. 90 ημέρες είναι η προβλεπόμενη περίοδος σε ένα σύνολο 180 ημερών και έχουμε και ένα παράρτημα στο οποίο εξηγούμε πώς γίνεται ο υπολογισμός των ημερών αυτών. Δεν εφαρμόζεται σε άτομα τα οποία ταξιδεύουν προκειμένου να απασχοληθούν κάπου στη συνέχεια, δηλαδή αυτούς που ψάχνουν εργασία και Υπάρχουν ξεχωριστέ κατηγορίες όσον αφορά αυτούς οι οποίοι ταξιδεύουν για επαγγελματικού λόγους αλλά δεν καλύπτονται αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν προς τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωση για να εργαστούν εκεί. Και κάτι ακόμα. εφαρμόζεται επίσης και στι συνδεδεμένε χώρε, όχι βάσει των συμφωνιών αυτών, αλλά λέμε ότι θα πρέπει να, έχουν, να συνάψουν οι χώρες αυτές με τις συνδεμένες με την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες διμερείς συμφωνίες. Και αυτό ισχύει και για τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία δεν εφαρμόζουν το κεκτημένο του Σέγγεν πλήρως. Ξέρετε ότι ε, δεν προβλέπεται τη δυνατότητα εισόδου στο χώρο Σέγγεν, πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένα κριτήρια αλλά επιτρέπεται για τους ανθρώπους αυτούς που θα υποφελούνται από την απαλλαγή αυτή θεώρησης να μπορούν να περάσουν για τη συγκεκριμένη αυτή περίοδο των 90 ημερών στο χώρο Σέγγεν. Πρέπει λοιπόν να τροποποιηθεί ανάλογο κανονισμός 539-2001 για τις χώρες αυτές. Ευχαριστώ. Στο μεταξύ κατεύθυνση και η φυγήτριά μας, η κυρία Μαρία Γκαμπριέλ. Ε, διαπραγματεύσεις στο τέλη του 2014 ήδη ξεκίνησαν για την άρση υποχρέωση θεωρήση διαβατηρίου και το Μάιο του 2015 υπεγράφησαν και τώρα έχουν έρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι προτάσεις προς ε, χωρίς σύμφωνης Μαρία, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα αρχίσω λέγοντας φυσικά ότι το θέμα αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ στο Κοινοβούλιο και μας είναι πολύ και με χαρά κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα να πω ότι πέρα από τη τεχνική διαδικασία έγκρισης που μα απασχολεί για κάθε μια από τι εκθέσει αυτέ, θα πρέπει να αξιολογήσουμε την πολιτική διάσταση ε, ε, της ε, από την υποχρέωση θεώρηση και για του δικού μα πολίτε και για την εξωτερική πολιτική τη Ένωση. Η σύναψη συμφωνιών με τρεις χώρες ΑΚΕ, ε, οχτώ χώρες ΑΚΕ που αναφέρατε προηγουμένω είναι πολύ σημαντική και εγγράφεται στη συνέχιση της εταιρική σχέσης που έχουμε στα πλαίσια της Συμφωνίας του Κοτονού, στην αναπτυξιακή μας συνεργασία, τον πολιτικό διάλογο και τους δεσμούς που έχουμε, ιστορικούς, ε, πολιτισμικούς και εμπορικούς. Επίσης, για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τονίζω ότι είναι η πρώτη αραβική χώρα που συνάπτει τέτοια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα πρέπει να εγγραφεί σε μια ευρύτερη ε, εικόνα, ε, συνεργασία των δύο χωρών που έχουν ε, κοινά συμφέροντα να σταθεροποιήσουν τη μακροπεριφέρεια και να είμαστε γεροί στη βαρύ και αξιόπιστη. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν ε, δεσμευτεί για πλήρη αμοιβαιότητα από το Μάρτιο του 2014 για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει συσταθεί και ομάδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά μπορούν να αποτελέσουν παραδείγματα για άλλες χώρες της περιοχής που θα επιθυμούσαν να συνάψουν τέτοια συμφωνία. Αυτή η συμφωνία απαλλαγής θεώρησης για βραχία διαμονή είναι ε, πραγματικά ένας ε, στόχος τον οποίο επιτύχαμε για να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας αλλά και ένα μέσο για να ε, συσφιχθούν έτσι περαιτέρω οικονομικές και εμπορικές σχέσεις και να εμβαθυνθεί ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες η απαλλαγή από τη θεώρηση ευατηρίου διανοίγει και οικονομικές ευκαιρίες και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις χώρες αυτές, είτε με αύξηση του τουρισμού, είτε με διευκόλυνση των ταξιδιών για επιχειρηματίες και επενδυτές. Και ακριβώς βλέπουμε στις χώρες αυτές ότι ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για τον τουρισμό και για να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους, η κάθε χώρα δηλαδή, αλλά και για άλλους λόγους. Και μας μας ενδιαφέρει πολύ και να πούμε ότι υπάρχουν χώρες όπου δεν υπάρχει κανένα προξενείο κράτους μέλους και για να ζητήσουν ε, βίζα Σέγγεν οι πολίτες της εν λόγω χώρας πρέπει να μεταβούν στο εξωτερικό, πράγμα που σημαίνει πλέον κόστος. Και για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ξέρουμε ότι η υποχρέωση θεώρηση, το κόστο θεώρηση, ο προγραμματισμό κτλ. είναι από τα βασικότερα εμπόδια για να πραγματοποιηθεί αυτό το ταξίδι. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι οι συμφωνίες αυτές θα πρέπει να μας χρησιμεύσουν ως εργαλείο για να φτάσουμε να επιτύχουμε τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής. 19 χώρες το 2014 με βάση ένα κανονισμό μεταφέρθηκαν στη ε, λίστα των ασφαλών κρατών και ε, αυτό συνεισέφερε θετικά στην όλη προσπάθεια. Στην έκθεσή μου θα επιμείνω στο να υπάρχει επαγρύπνηση και αυστηρή παρακολούθηση και μετά τη σύναψη των συμφωνιών ε, παρακολούθηση είτε των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είτε τη στήριξη τη αρχή της αμοιβαιότητα. Παρά το γεγονό ότι δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για τις χώρε αυτές, είναι χαμηλή σήμερα η ε, άρνηση, ή μάλλον το ποσοστό απόρριψη για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα επίσης και αυτό δείχνει ότι υπάρχει εμπιστοσύνη απέναντι στους πολίτες των χωρών αυτών. Βέβαια, ως συγκήτρια θα ήθελα να ζητήσω και εγώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποιες διευκρινήσεις μετά από αυτά τα εισαγωγικά που είπα. Θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας μιλήσει λίγο περισσότερο για την ασφάλεια των ταξιδιωτικών εγγράφων των διαβατηρίων και επίσης πώς γίνεται να αποτραπεί η ε, απόκτηση της ηθαγένειας της ε, εν λόγω χώρες για να διευκολυνθούν τα ταξίδια προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, βλέπε δομινικά. Λυπάμαι που το Κοινοβούλιο δεν ενημερώνεται εγκαίρως για την πρόοδο των διμερών διαπραγματεύσεων. Το 2014 μεταφέραμε λοιπόν 19 χώρες το θετικό κατάλογο και δράτω με τις ευκαιρίες για να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι γίνεται με τις διαπραγματεύσεις με τις 10 υπόλοιπες χώρες, εκ των οποίων 8 είναι χώρες ΑΚΕ. Ε, Προηγουμένω μίλησα για τα κριτήρια μετά την σύναψη συμφωνία και πώ τα παρακολουθούμε. Και επειδή εμεί είμαστε άμεσα εκλεγμένο όργανο και είμαστε και υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια μεικτή επιτροπή. Το είπα από πέρσι και το τόνισα και το έθεσα υπόψη σας. Ποιος ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη μεικτή Επιτροπή Διαχείρισης αυτών των συμφωνιών. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διαδραματίζει ένα ρόλο πιο πρωταγωνιστικό. Και τι γίνεται με την προσωρινή εφαρμογή των συμφωνιών πριν την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για ποιο λόγο αυτό, τι το δικαιολογεί. Κατανοώ ότι θέλετε να μειώσετε τις διαδικασίες που καμιά φορά είναι πολύ περίπλοκες και χρονοβόρες για τις χώρες και θέλετε οι εξαιρέσεις και οι απαλλαγές να τεθούν σε ισχύ το συντομότερο. Αλλά εάν το Κοινοβούλιο εμπλεκόταν περισσότερο και πιο στενά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, Είμαι πεπισμένη ότι θα φτάναμε στο ίδιο αποτέλεσμα χωρίς να περιορίζεται το περιθώριο ελιγμών και χειρισμών του Κοινοβουλίου στην απόφαση του. Και έχω και ερωτήσεις για τις ε, συμφωνίες που ήδη εφαρμόζονται από το Μάιο. Έχει ήδη στοιχεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κινητικότητα των πολιτών αυτών των χωρών προς την Ένωση και τούμπαλη. Συμπεραίνω λέγοντας ότι ε, ως εισηγήτρια χαίρομαι πάρα πολύ ε, για την πρόταση αυτή. Είμαι υπέρ του να το δώσει τη θετική του γνώμη το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ τους και εισηγητές και τα μέλη της Επιτροπής μας που καλό να εκφράσουν τη γνώμη τους και θα ήθελα εκ των προτέρων να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις απαντήσεις και για τη συνεισφορά της για να μπορέσει το Κοινοβούλιο το συντομότερο να δώσει τη θέση του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητή Μαρία Γκάμπριελ, η Άννα Γκόμες. Χαίρομαι πολύ που βλέπω τη Μαρία ξανά πίσω στο κοινοβούλιο. Θα σας διαβάσω τις ε, σημειώσεις της Σιλβίγκη Γιώμα, που είναι σκιώδης, η οποία ακριβώς λέει αρχικά στις σημειώσεις της ότι λυπάται που δεν μπορεί να είναι εδώ στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων για αυτές τις συμφωνίες. Ίσως και να μην είναι χρήσιμο να το επενθυμίσουμε, αλλά η πολιτική των θεωρήσεων και οι συμφωνίες ε, τύπος που μελετούμε είναι πολύ σημαντικές για να έχουμε περισσότερη κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταξύ Ένωσης και τρίτων χωρών γιατί επίσης συνεισφέρει και στην εμβάθυνση, τη μεγαλύτερη εμβάθυνση των σχέσεων της Ένωσης με τις τρίτες χώρες. Ε, Πρόκειται για μια ανανομένη συνεργασία που θα επηρεάσει την κινητικότητα αλλά και άλλες σημαντικές πτυχές όπως είναι η ανάπτυξη της, ε, των πολιτιστικών, ε, κοινωνικών, οικονομικών και άλλων δεσμών, ενισχύει τις επαφές μεταξύ των λαών, ε, και συγκεκριμενοποιεί και την ελευθερία της κυκλοφορίας που είναι θεμελιώδες δικαίωμα στην Ένωση. Σε αυτή τη φάση επομένω θα ήθελα πολύ συγκεκριμένα τρία στοιχεία να τονίσω. Πρώτον, την ανάγκη υλοποίηση ενός μηχανισμού αμοιβαιότητας. Δεύτερον, τη σημασία να παρακολουθεί το Κοινοβούλιο την εφαρμογή αυτών των συμφωνιών, άρα την ανάγκη να τηρείται ενήμερο τακτικά και πλήρως σε σχέση με την εφαρμογή των συμφωνιών όπως προβλέπει η αρχή της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Και τρίτον, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το θέμα αυτό χρήζει ιδιαίτερη προσοχή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπογραμμίζει η Σιλβή ότι χαίρεται πολύ ε, και περιμένει ότι θα υπάρξει πολύ επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων με την Μαρία και τους άλλους ε, σκιώδεις. Κολεγίν Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ με τη σειρά μου να πω ότι χαίρομαι πολύ που ξαναβλέπω τη Μαρία μεταξύ μας. Είναι μεγάλη χαρά να συνεργαζόμαστε. Χαίρομαι πολύ λοιπόν ε, είμαι εγώ εκπεπτήσως υπέρ της απελευθέρωσης ε, των θεωρήσεων βραχίας διαμονής. Θα δείτε και από ε, τις μελέτες που έχουν γίνει ότι αυτές οι θεωρήσεις βραχίας διαμονής δημιουργούν πιο πολλά προβλήματα από αυτά που λύνουν. Άρα, επειδή δεν έχω κάποιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Συμφωνώ με τις προκαταρκτικές παρατηρήσεις και της Μαρία και της Σιλβίδια Στόματος Αναγκόμες Βέβαια με ενοχλεί κάπω που ουσιαστικά επιλαμβανόμαστε εκ των υστέρων του θέματος. Οι συμφωνίες εφαρμόζονται ήδη. Άρα είμαστε πρωτοτελεσμένοι. Δεν είναι καλό αυτό. Όποιοι και αν είναι λόγοι, δεν ήταν τόσο πια κατεπήγον, ώστε να μην δοθεί η πρώτερη έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν ξέρω, μήπως ε, επειδή είναι πριν το καλοκαίρι, και είναι τουριστικοί λόγοι πάνω απ' όλα για την απελευθέρωση, γιατί αν έχουν κάτι κοινό αυτέ οι χώρε είναι ότι είναι τουριστικοί προορισμοί για επικόστον των χωρών μα. Να κάνω και μια παρατήρηση για τη λογική του πακέτου. Γιατί ένα πακέτο πέντε από τι ε, χώρες Καραϊβικής, δύο Νότιου Ειρηνικού και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυρά. Εκεί έχω και ακόμα περισσότερα ερωτηματικά, δεν είναι και τόσο τουριστικός προορισμός, εσείς μετά άλλο άλλα τουλάχιστον κράτη. Χαίρομαι πάντως που υπάρχει η αρχή της αμοιβαιότητας στο κέντρο των συμφωνιών. Αυτή είναι η αρχή που πρέπει να μας καθοδηγεί ε, πάντοτε, αλλιώς δεν είναι κατανοητό προς τα έξω. Να κάνω και μια πιο γενική παρατήρηση. Για τις πρεσβείες. Το έθεσε η Μαρία το θέμα. Είναι και αυτό το επίκεντρο της μέτρων για τι θεωρήσει. Ελπίζω γρήγορα να έχουμε τα δύο σχέδια έκθεσης για τη δέσμη μέτρων για τη θεωρήσει. Το ένα καθυστερεί η μία έκθεση ε, και θα ήθελα να γνωρίζω γιατί καθυστερεί τόσο πολύ από του δύο εισηγητές. Ποια είναι τα κινητρά του. Αυτά και ευχαριστώ για μια ακόμη φορά τη Μαρία και προσβλέπω στη μεταξύ μας συνεργασία έχουμε ραντεβού νομίζω το Σεπτέμβρη για να επεξεργαστούμε πιο δεξοδικά όλες αυτές τις προτάσεις. Αλλά ε, συνοψίζοντας είμαι θετικά διακείμενη στις προτάσεις αυτές. Τι είναι εξαιρετικό. Επόμενη συνάδελφος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μιλάω τη γλώσσα μου, τα ειδικά. φορέστε λοιπόν τα ακουστικά σας, σας παρακαλώ. Νομίζω ότι όσο περισσότερες απαλλαγές έχουμε από την υποχρέωση θεώρησης, τόσο το καλύτερο. Πρέπει να επιτρέπουμε στους πολίτες αυτούς και τους δικούς μας και των άλλων χωρών να κυκλοφορούν ελεύθερα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι θετικό το ότι εγκρίνουμε αυτές τις συμφωνίες. Άκουσα ότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα όσον αφορά το ζήτημα της ηθαγένειας. Άρα νομίζω ότι η συγγήτρια απάντησε και σε αυτά. Τι γίνεται όμως τώρα με τη συγκεκριμένη συμφωνία. Και όσον αφορά τα Ενωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ξέρετε ότι έχουμε καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά ελπίζω ότι θα αλλάξει η κατάσταση και ότι θα αρχίσουν να σέβονται περισσότερο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καταλαβαίνετε ότι δεν προασπίζονται παρκώς τα ανθρώπινα δικαιώματα στις χώρες αυτές. Είναι πολύ θετικό το ότι έχουμε όλα αυτά τα μέτρα διευκόλυνσης των θεωρήσεων. Απαιτείται αυτό το πράγμα και νομίζω ότι υπάρχουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι και πολλές φορές άνθρωποι προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα ή εργάζονται για μη κυβερνητικέ οργανώσει που προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν ανάγκη τις θεωρήσεις αυτές για να ταξιδεύουν πιο εύκολα ή μάλλον τα συστήματα αυτά κατάργησης της υποχρέωσης θεώρησης. Ευχαριστώ πολύ. Η συνάδελφος Κέγκε, η συναδελφος παρακαλω Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ με τη σειρά μου χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναβλέπω τη Μαρία. Το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι ασχολούμεθα πολύ με το ζήτημα αυτό έχουμε όλες αυτές τις συμφωνίες εξαίρεσης από την υποχρέωση θεώρησης. Ξέρετε ότι εγώ συμμετέχω και στην αντιπροσωπεία και όπου ερχόμαστε σε επαφές με ανθρώπους οι οποίοι πολλές φορές ταπεινώνονται πραγματικά στην αντιμετώπιση που έχουν στις αιτήσει που κάνουν προκειμένου να φτάσουν εδώ πέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ταξιδέψουν και πολλές φορές ακόμα να συμμετέχουν στις δικές μας τις συναντήσεις. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως θεσμοί να αντιμετωπίσουμε τους ανθρώπους αυτούς με αξιοπρέπεια. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να εγκρίνουμε τις συμφωνίες αυτές και θα πρέπει να διέπονται βέβαια από διαφάνεια και από ισότιμη αντιμετώπιση όλων. Ξέρετε ότι μπορούν να συμβάλλουν περισσότερο στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και στον τουρισμό οι συμφωνίες αυτές. Και βέβαια θα διευκολύνουν και τις επαφές που έχουμε με τις χώρες αυτές. Θα μπορούσαμε όμως να λάβουμε υπόψη μας όλες τις χώρες εκείνες με τις οποίες έχουμε επίσημες σχέσεις, όπως για παράδειγμα τις υπόλοιπες χώρες ΑΚΕ. Ξέρετε ότι πάρα πολλέ φορέ εκπρόσωποι των χωρών ΑΚΕ περιμένουν πλέον μια θετική κίνηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω ότι η Μαρία έχει ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό, αλλά θα ήθελα και μια επίσημη απάντηση για να γνωρίσω τελικά πού βρισκόμαστε και αν τελικά προτιθέμεθα να εντάξουμε στου καταλόγου αυτούς και άλλες χώρες πέρα από αυτές που έχουμε στη συγκεκριμένη πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία πάσα μας έδωσε η κυρία Κιέγγι, διότι το λόγο έχει αμέσω τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you, Madam. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ορισμένες από τις ερωτήσεις της έθεσε η συγγήτρια ε, και άλλοι συναδελφοί σας ό,τι αφορά την ε, ασφάλεια των ταξιδιωτικών εγγράφων. Έχουμε την πρόταση του 12. Ε, πραγματικά με τις χώρες της Καραϊβικής εκτιμήσαμε ότι υπήρχε ε, υψηλό επίπεδο ασφαλείας των ταξιτικών εγγράφων της Καραϊβικής Κάρικομ, το ίδιο και για τα νησιά του Ειρηνικού που είναι αναγνώσιμα από μηχάνημα τα διαβατήρια αλλά δεν αποτελεί βιομετρικό, το βιομετρικό διαβατήριο προϋπόθεση για απαλλαγή από την ε, υποχρέωση θεώρησης. Θεωρήσαμε όμως ότι είναι επαρκής ε, προϋποθέσεις ασφάλειας. Τώρα πρόσβαση για πολίτες των χωρών. Υπάρχει το ζήτημα της λαθρομετανάστευσης, παράτυπης μετανάστευσης, υπάρχουν τα θέματα ασφαλείας, ε, αναλογίες, τα ποσοστά ε, επιστροφών κτλ θα τα αξιολογήσουμε όλα αυτά. Σε ό,τι αφορά πληροφορίες για τις άλλες χώρες, να πω ότι οι συμφωνίες με Περού και Κολομβία ξεκίνησαν τον Ιούνιο στα περιθώρια της ΕΛΑΚ και τώρα προετοιμάζουμε τις αστερικές διαδικασίες, ίσως οι υπογραφές να πέσουν το φθινόπωρο. Για Τόγκα, Κυρινάτη, Μαλάουι ξεκίνησαν διαδικασίες για τη μονογραφή και εκεί που δεν έχουμε ξεκινήσει έχουμε τα νησιά του Σολομόντα, Ναουρό, του Βαλού, Μικρονησία και νήσι Μάρσαλ. Για άλλα θέματα. Είπαμε ότι περάσαν και τέθησαν προσωρινά σε ισχύ σε διαφορετικές ημερομηνίες το Μάιο, πολύ πρόσφατα, 6 Μαΐου για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, 28 Μαΐου για την Καραϊβική, Σαμόα, Βανουάτου και 26 Μαΐου για το Τιμόρ Λέστε. Δεν έχουμε άλλα στοιχεία για αριθμούς, νούμερα, δηλαδή ποιοι ε, και πώς έχουν ταξιδέψει από αυτό το καθεστώς. Η Επιτροπή που θα διαχειρίζεται τις συμφωνίες. Το λένε στις συμφωνίες ότι η Ένωση εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή τη Διεχειριστική Επιτροπή που δεν συνέρχεται συχνά, δεν είναι το ίδιο με τις συμφωνίες ε, για την διευκόλυνση ε, χωρίς θεώρηση διαβατηρίου. Εδώ είναι κάτι διαφορετικό, υπάρχει αμοιβαιότητα, αλλά όπως λέγεται και στη συμφωνία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκπροσωπεί σε περίπτωση που χρειαστεί σε αυτή τη Διεχειριστική Επιτροπή την Ένωση. Για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ένα ερώτημα. Δεν ήταν στην πρόταση της Κομισιόν, αλλά οι συνομοθέτες το προσέθεσαν σε διαπραγματεύσεις. Η ΕΕΔ αξιολόγησε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα και τώρα κατά πόσον υπάρχουν και άλλες χώρες που στο μέλλον μπορεί να μπουν σε αυτό το καθεστώς. Να σας υπενθυμίσω ότι η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι μέχρι τα τέλη του έτου θα καταθέσει πρόταση για μεταφορά από το θετικό στον αρνητικό κατάλογο λόγω ε, κάποιων χωρών ή το αντίστροφο και θα την έχετε μέχρι τα τέλη του χρόνου αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφόρηση. Μαρία, θέλεις να ξαναμιλήσεις? Ναι, μόνο να πω ότι θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους συναδέλφους για τα όσα είπαν και το Σεπτέμβριο όντως θα συνεδριάσουμε με τους συγκεκριτές και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Α, η κυρία Βερζιά έχει ερώτηση. Ναι, ζητώ συγγνώμη. Αλλά θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας εφώτισε. Θα ήθελα λίγο πιο συγκεκριμένες απαντήσεις για τις προσωρινές συμφωνίες και είπατε, απαντώντας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι αξιολογήθηκαν ε, μπορούμε να έχουμε αυτές τις αξιολογήσεις γιατί θα μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Ήταν ενδιαφέρουσες. Θέλετε να απαντήσετε και πάλι πρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ναι, ίσως για αυτό το θέμα που έχει να κάνει με αυτή την ερώτηση. Ε, δεν ήταν ε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αρχικά στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γι' αυτό έγινε αξιολόγηση Υπάρχει ένας διάλογος ε, με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης με τα ε, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα όπου συζητούν και τέτοια θέματα. Αυτή είναι η αξιολόγηση, όχι από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εντάξει, δεν θα πρόκειται να λύσουμε εμείς αυτά τα προβλήματα συνολικά, θα βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας. Ευχαριστώ πολύ. Tagesordnungspunkt, nämlich Tagesordnungspunkt 30. Ευχαριστώ. Προχωρούμε στο σημείο 30, παρουσίαση των ε, διάμεσων εκθέσεων από το θεματικό τμήμα για τα δικαιώματα των πολιτών και τις συνταγματικές υποθέσεις. Έχουμε ε, αναθέσει τις εξή εκθέσεις και μελέτες. Πρώτον, ενίσχυση του κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου και εναλλακτικέ λύσεις στη Συμφωνία του Δουβλίνου. Καλωσορίζω ε, τους εμπειρογνώμονες και ε, χαίρομαι που ε, είναι κάθοδον προς το πάνελ και τους προσκαλώ στο Προεδρείο για να μας κάνουν μια σύντομη παρουσίαση της πρώτης μελέτης. Ε, στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες στον τομέα της μετανάστευσης και τέλος η τρίτη μελέτη μας είναι η εξερεύνηση νέων οδών όσον αφορά την νομοθεσία για τη μετανάστευση για λόγους εργασίας και την οικονομική μετανάστευση. Legale Arbeits- und Wirtschaftsmigration befassen. Αυτά λοιπόν, αυτές είναι τρεις εκθέσεις. Ευχαριστώ τις δύο κυρίες που ήρθαν σε αυτή την προκεχωρημένη ώρα. Είναι το τελευταίο θέμα μας πριν στις ειρηνές διακοπές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Θα δώσω μέσα στο λόγο στις δύο κυρίες, κυρία Γκίλτ και κυρία Γκάλικ. Έχετε 10 λεπτά για όλη τη μελέτη και οι δυο σας. Έχετε μέσα στο λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Very Σας ευχαριστώ πολύ. Ιδιαίτερη ευχαρίστηση να βρίσκομαι στην Επιτροπή σας Έχουμε κάνει μια πολύ λεπτομερή μελέτη, η οποία πολύ σύντομα πρόκειται να δημοσιευθεί για την ενίσχυση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και για την εξέβρεση εναλλακτικών λύσεων στη Συμφωνία του Δουβλίνου όσον αφορά την κατανομή των ετούντων άσυλο. Το πρώτο ζήτημα λοιπόν το οποίο τίθεται και το οποίο μελετήσαμε μετά την ε, μελέτη που προετοιμάσαμε για σας και σας παρουσιάσαμε το Δεκέμβριο, ήταν πώς το σύστημα του Δουβλίνου μπορεί να συμβάλλει ή πώς συμβάλλει στις μη ασφαλείς αφήξεις προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαντώντας λοιπόν το ερώτημα αυτό, η μελέτη μας επικεντρώνεται στο πώς πολλές φορές ε, λειτουργεί η γνώση αλλά και ο φόβος του συστήματος του διβλούνιου από τους ετούντες άσυλο ή τους πρόσφυγες, ότι πολλές φορές ουσιαστικά προσπαθούν να αποφύγουν οποιαδήποτε επαφή με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών προορισμού ή των κρατών μελών από τα οποία περνούν και μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί φοβούνται ότι πρόκειται να τους επιβληθούν συγκεκριμένα μέτρα που πολλές φορές έχουμε ουσιαστικά επιστροφή, ακόμα και στην περίπτωση της Ελλάδας. Το επόμενο, το ερώτημα το οποίο θέσαμε, πάντα σε σχέση με τις μη ασφαλείς και επικίνδυνες αφήξεις ε, των άσυλων και προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ποια είναι τα εμπόδια όσον αφορά την ασφαλή είσοδο των προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δείτε ότι στην έκθεσή μας προσπαθήσαμε να δούμε ποιος τελικά φτάνει ασφαλώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό συνάδει πολύ με τη συζήτηση που μόλις κάνατε όσον αφορά τις απαιτήσει χορήγηση θεώρηση. άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη από θεώρηση φτάνουν τελικά ασφαλώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούν να πάρουν από την Τίνιδα ένα ferry boat, να φτάσουν στην Ιταλία για 35 μόνο ευρώ και συνέχεια μπορούν να πάρουν μια πτήση από την Ιορδανία μέχρι το Παρίσι για 300 περίπου ευρώ. Και προφανώς δεν χάνουν τη ζωή τους διασχίζοντας τη Μεσόγειο έχοντας ε, καταβάλει σύμφωνα με τα δεδομένα του UNCHR 5 με 7.000 δολάρια για να μη ασφαλές προφανώς ταξίδι. Ποια είναι λοιπόν τα μέσα τα οποία είναι διαθέσιμα όσον αφορά τις ασφαλείς αφήξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δούμε ποια είναι τα εμπόδια καταρχάς. Το πρώτο εμπόδιο είναι η υποχρέωση θεώρησης. Το δεύτερο εμπόδιο είναι οι κυρώσεις απέναντι στους διακινητές και κυρώσει μάλλον για τις εταιρείε μεταφοράς οι οποίοι μεταφέρουν ενδεχομένως ανθρώπους χωρίς να έχουν τα απαραίτητα ταξιωτικά έγγραφα. Και πρέπει λοιπόν να δούμε ακριβώς τι προβλέπεται για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι πρέπει να έχουν θεώρηση και αν δούμε τις δέκα πρώτε, χώρε πρώτες χώρες ετούντων άσυλων βλέπουμε ότι υπάρχει μόνο μία χώρα για την οποία δεν απαιτείται θεώρηση και αυτή είναι η Σερβία. Ποιους μηχανισμούς λοιπόν θα, μπορέσ, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να εξασφαλίσουμε ασφαλή είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα, μπορέσουμε, θα μπορούσαμε να καταργήσουμε την υποχρέωση θεώρησης, αυτό το οποίο συζητήσατε μόλις πριν από λίγο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει δραστηριοποιηθεί στην Ανθρωπιστική Εκένωση για τους δικούς τους πολίτες αλλά και για πολίτες τρίτων χωρών. Επίσης έχουμε προετοιμάσει μία μελέτη για σας πριν από ένα χρόνο σχετικά αφορά το ζήτημα των ανθρωπιστικών θεωρήσεων και πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Και έχουμε τα παραδείγματα κάποιων κρατών μελών που ήδη δίνουν τέτοιες ανθρωπιστικές θεωρήσεις. Και έπειτα Έχουμε και το ζήτημα των υφιστάμενων μεταναστευτικών διαδρομών. Αν δούμε τους ετούντες άσυλο από χώρες όπου μάλλον υπάρχουν πολλοί ετούντες άσυλο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε ότι οι χώρες αυτές υπόκεινται στην απέτηση θεώρησης. Για παράδειγμα, αν πάρουμε τη Συρία και το Ιράκ, συνειδητοποιούμε ότι πάρα πολλοί πολίτες τους ακολουθούν κάποιους μη ασφαλείς δρόμους, οδούς, προκειμένου να φτάσουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές φορές ταξιδεύουν με σκάφη, αλλά προφανώς οι Ουκρανοί ακολουθούν άλλους δρόμους, οι οποίοι είναι πιο ασφαλείς. Όταν οι Ρακινοί οι Σύριοι προσπαθούν να περάσουν από την Τουρκία στην Ελλάδα ή προς τη Βουλγαρία, πάλι με στοιχεία του UNCHR και από την Human Rights Watch, βλέπουμε ότι οι πολίτες αυτοί αντιμετωπίσουν τακτικές ακραίας βίας που έχουν οδηγήσει πολλές φορές στο θάνατο ορισμένων πολιτών, επομένω αποθαρρύνονται από το να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πιο ασφαλεί οδού. Μα ζητήθηκε επίσης στα πλαίσια της μελέτης αυτής να δούμε τι γίνεται με τα κέντρα υποδοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σε υπενθυμίσουμε ότι Σύμφωνα με το Άμεθ και το Ταμείο για τους Πρόσφυγες, αυτά τα κέντρα υποδοχής αλλά και οι συνθήκες υποδοχής εκεί πέρα χρηματοδοτούνται πολλές φορές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτά τα κέντρα υποδοχής ουσιαστικά σε οποιοδήποτε κράτος μέλος και βρίσκονται είναι κέντρα υποδοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας ενοχλεί πάρα πολύ το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται πολλές φορές μέτρα καταστολής κατά των ε, ετούν τον άσυλο κατά των προσφύγων και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πληρούνται όλες οι συνθήκες σωστής υποδοχής σε όλα αυτά τα κέντρα υποδοχής σύμφωνα με τη σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα ζητήθηκε επίσης να εξετάσουμε και τα κέντρα υποδοχής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να επιστήσουμε εδώ πέρα την προσοχή σας στο ότι υπάρχουν πάρα πολλά επιχειρήματα τα οποία τα αναφέρουμε και στην έκθεσή μας και γενικά θεωρείται ότι αυτά τα κέντρα υποδοχής από πάρα πολλές τρίτες σε τρίτε μάλλον χώρε, δεν είναι αποτελεσματικά και γενικά δεν ενδείκνυται. Να περάσουμε τώρα στο δεύτερο τμήμα της έκθεσης αυτής. Αν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης όσον αφορά τις θετικές αποφάσεις χορήγησης ασύλου. Ξέρετε ότι οι αρνητικές αποφάσεις αυτή τη στιγμή αναγνωρίζονται από τον κανονισμό του Δουβλίνου και στην περίπτωση αυτή πρέπει κανείς να επιστρέψει στη χώρα προέλευσης και όλες αυτές οι αποφάσεις εφαρμόζονται στα πλαίσια των αποφάσεων επιστροφής. Πρέπει όμως να δούμε τι θα γίνει και με τις θετικές αποφάσεις, δηλαδή αυτές που χορηγούν τελικά άσυλο. Και ξέρετε ότι σε πάρα πολλέ νομοθεσίε Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τι εσωτερικέ υποθέσει στη δικαιοσύνη προβλέπεται μια αμοιβαία αναγνώριση συγκεκριμένων αποφάσεων. Νομίζω πάντως ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει απαραίτητη εναρμόνιση στον τομέα του ασύλου. Η ε, αμοιβαία λοιπόν αυτή αναγνώριση των θετικών αποφάσεων χορήγησης ασύλου απορρέει τελικά από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκής Ένωση και συγκεκριμένα από το άρθρο 78 που αποτελεί τη νομική βάση για μια κοινή πολιτική για το άσυλο προκειμένου να υπάρχει το κατάλληλο καθεστώς για όλους εκείνους οι οποίοι χρήζουν διεθνούς προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συνάδει και με την ε, Σύμβαση της Γενέβης. Πρέπει λοιπόν να υιοθετηθούν μέτρα προκειμένου να έχουμε ένα κοινό σύστημα ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο να περιλαμβάνει ένα ομοιόμορφο καθεστώς για τους ετούντες άσυλο που να παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων λοιπόν που λαμβάνονται από τα μεμονωμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να ενισχύσουμε την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου όπου θα πρέπει να τηρούνται και τα θεμελιώδη δικαιώματα και η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας και θα μπορέσουμε να κάνουμε και επενδύσεις στην οικοδόμηση ικανοτήτων στα κράτη-μέλη, ιδίως στα κράτη-μέλη αυτά που υστερούν και δεν έχουν ακόμα συμμορφωθεί με την κοινοτική νομοθεσία και που δεν έχουν εναρμόσει ουσιαστικά την νομοθεσία τους. Και επίσης κατά αυτόν τον τρόπο θα μετριάσουμε και τις αρνητικές επιπτώσεις του συστήματος του Δουβλίνου, όπου πολύ συχνά βλέπουμε ότι οι αρμόδιες αρχές σε ένα κράτος μέλος όσον αφορά τη χορήγηση ασύλου είναι επίσης οι αρμόδιες αρχές για την διεθνή προστασία για μια περίοδο πέντε ετών. Και βλέπουμε ότι ε, στις ε, περιπτώσεις αυτές, όταν δηλαδή η ίδια αρμόδια αρχή ασχολείται τόσο με τη διεθνή προστασία όσο και το άσυλο, μπορεί ορισμένοι πολίτες σε περίπτωση άρνηση του ενός να μην καταφέρουν καν να εξασφαλίσουν ούτε το δεύτερο καθεστώς. Στην έκθεση αυτή λοιπόν εξετάζουμε δύο εναλλακτικέ όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση στο κοινοτικό δίκαιο. Η πρώτη εναλλακτική που περιλαμβάνει μια αμοιβαία αυτόματη αναγνώριση του καθεστώτος του ετούντος άσυλο και η δεύτερη εναλλακτική που προβλέπει το καθεστώς προστασίας του προσφύγου από την πρώτη μέρα που θα πρέπει να ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε και ένα καθεστώς ελεύθερης ε, κυκλοφορίας για αυτούς τους ανθρώπους. και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε τελικά να πετύχουμε και τους στόχους της συνθήκης. Αλλά ενδεχομένως εδώ πέρα να ελοχεύει ο κίνδυνος να μην μπορέσουμε τελικά να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο λέμε ότι η σύσταση αυτή μαζί με κάποιες άλλες συστάσεις που γίνονται στη μελέτη αυτή, θα πρέπει να συνοδεύονται από περισσότερες προσπάθειες για την εφαρμογή των υφιστάμενων υποχρεώσεων για το άσυλο παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δεύτερη εναλλακτική που προβλέπετε εδώ και την οποία σας προτείνουμε, είναι μία η οποία θα περιλαμβάνει λιγότερες αλλαγές στο φυστάμενο νομικό πλαίσιο, δηλαδή συντόμευση της περίοδου μετά την οποία μπορεί να δοθεί σε κάποιον προστασία και όπου θα μπορεί να μεταβαίνει σε ένα άλλο κράτος μέλος. Από τα πέντε χρόνια που έχουμε αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να περάσουμε σε μια περίοδο δύο ετών. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να πάνε ορισμένοι πολίτες σε κάποια άλλα κράτη-μέλη, στα οποία ενδεχομένω να ενσωματώνονται πιο γρήγορα και καλύτερα. Παράλληλα όμως, οι πολίτες αυτές θα αναγκάζονται να ενσωματωθούν περισσότερο στις χώρες εκείνες που τους παρέχουν προστασία. Σύμφωνα με μια τέτοια διάταξη θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε τις προϋποθέσεις που υφίστανται αυτή τη στιγμή όσον αφορά τη δυνατότητα μετακίνησης σε άλλη χώρα με συγκεκριμένε εξαιρέσεις όσον αφορά τις ε, περιπτώσεις ανθρωπιστικών κρίσεων. Στη συνέχεια αναφερόμαστε σε κάποιες εναλλακτικέ όσον αφορά την ίδια τις, τις ίδιες τις διατάξεις του Δουβλίνου και προβλέπουμε πάλι εδώ πέρα κάποιες ε, εναλλακτικέ. Λέμε ότι θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό οργανισμό για τη μετανάστευση, το άσυλο και την προστασία. Δηλαδή ένα οργανισμό ο οποίος θα μπορούσε πραγματικά να, να επεξεργάζεται όλες τις αιτήσει ασύλου, οπουδήποτε και αν υποβάλλονται αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μπορούσε να εξυπηρετεί όλα τα κράτη-μέλη βάσει συγκεκριμένων προποθέσεων που θα έχουν ήδη αποφασιστεί στα πλαίσια του νησιακού δικαίου. Η δεύτερη εναλλακτική είναι το να δώσουμε σε κάποιους πολίτες την δυνατότητα να επιλέξουν αυτοί που θέλουν να τηθούν διεθνούς προστασίας. Δεν είναι όμως ιδιαίτερα δημοφιλής η λύση αυτή με κάποια κράτη-μέλη και δεν νομίζουμε ότι με το εφιστάμενο πολιτικό πλαίσιο θα εγκριθεί. Θα μπορούσαμε στη συνέχεια να έχουμε ένα σύστημα επανατοποθέτησης των προσφύγων μετά την αναγνώριση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας και μια τέταρτη εναλλακτική θα ήταν η επαντοποθέτηση των ετούντων άσυλο σε άλλα κράτη-μέλη βάσει μιας κλίδας κατανομής που θα λαμβάνει υπόψη της ε, τον πληθυσμό της χώρας, την οικονομική ανάπτυξη της χώρας καθώς επίσης και τις σχέσεις που ενδεχομένω η χώρα αυτή να έχει, η χώρα προορισμού με τη χώρα προέλευσης. Στο τέλος της μελέτης αυτής προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση, τη χρηματοδοτική συνδρομή προς τις χώρες εκείνες οι οποίες δέχονται ιδιαίτερη πίεση, χώρες οι οποίες δεν μπορούν να αποκριθούν τις υποχρεώσεις τους. Μια επιλογή που θα ήταν η πιο εύκολη από νομικής πλευράς θα ήταν να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση, της χρηματοδότησης στα πλαίσια του Ταμείου Μετανάστευσης Ασύλου και ενσωμάτωση. Ξέρετε ότι ήδη έχουν αυξηθεί τα κονδύλια του Ταμείου αυτού σε σχέση με την προηγούμενη ε, περίοδο προγραμματισμού, αλλά λαμβάντα υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις βλέπουμε ότι και πάλι η αύξηση των κονδυλίων δεν αρκεί για να καλυφθούν οι ανάγκες, ιδίως στις χώρες εκείνες που δέχονται περισσότερη πίεση. Μία δεύτερη δυνατότητα θα ήταν να δημιουργηθεί ένα συγκεκριμένο ταμείο στα πλαίσια του κοινοτικού προπολογισμού, ταμείο το οποίο θα έχει ως στόχο να διασφαλίσει περισσότερη αλληλεγγύη στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την άνηση αυτή ε, οικονομική πίεση που ε, ασκείται σε ορισμένε χώρες εξαιτία τη μετανάστευση. Σε κάθε πάντω περίπτωση θεωρούμε ότι η χρηματοδότηση πρέπει να αυξηθεί και θα πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένα μέτρα όπου να, να, δέχονται, να τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι καθώς επίσης και δείκτες συγκριτική αξιολόγηση για την πιο αποτελεσματική χρησιμοποίηση αυτών των κονδυλίων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπατε στο τέλος, ότι το πιο απλό θα ήταν περισσότερα χρήματα. Εγώ είμαι μέλο τη επιτροπή προπολογισμών και έχω απέναντί μου διαφόρου που δεν είναι και τόσο κυμπάριδε. Να δούμε λοιπόν πώ θα τα χειριστούμε αυτά τα θέματα. Ξέρετε, έχουμε ήδη πρόβλημα χρόνου, δεν ξέρω αν έχουμε ερωτήσει, οι συνάδελφοι. Η κυρία Γκόμες. Uh, Σύντομα θέλω να πω ότι αυτό το θέμα της χρηματοδοτικής υποστήριξης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ γνωρίζω στη χώρα μου που είναι μία από τις χώρες που δέχεται τους λιγότερους πρόσφυγες διότι δεν έρχονται στην Πορτογαλία ε, όσοι έρχονται στις άλλες χώρες. Ξέρω τι συμβαίνει για διάφορους λόγους, σε πάση περιπτώσει, δεν έρχονται στην Πορτογαλία, αλλά ξέρω δημάρχους από περιοχές της υπέρθρου που έχουν απεριμωθεί λόγω της αστιφιλίας στην αρχή και της οικονομικής κρίσης στη συνέχεια. 485.000 άνθρωποι έχουν μεταναστεύσει την τελευταία τετραετία και ξέρω λοιπόν ότι υπάρχουν δήμαρχοι που θα ήθελαν να υποδεχθούν ε, για μετεγκατάσταση πρόσφυγες, ανθρώπους που έχουν ανάγκη ή και μετανάστες, εργάτες, υπό την προϋπόθεση ότι θα είχαν τη σωστή οικονομική υποστήριξη για να τους εγκαταστήσουν όπου, σε περιοχές όπου υπάρχουν ε, ε και προς ακόμα και σπίτια για να τους στεγάσουν. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να δούμε και να το πιέσουμε και να δοθεί ως κίνητρο. Ε, actually, accept. <laughs> για να μπορέσει ε, να ε, γίνει αποδεκτή αυτή η κλίδα να διανομήσει. κυρία Βεζιά ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα κυρίως να σας ευχαριστήσω κυρίες μου για την έκθεση αυτή. πολλές από τις συστάσεις σας πραγματικά ε, συμφωνούν, δικαιολογούν και τροφοδοτούν πολλές από τις δικές μας προτάσεις, γιατί είμαστε αρκετοί που συμφωνούμε. Δεν ξέρω, ίσως χαριτολογώντας να πω και στη σχέση με τα όσα είπε η κυρία Χολμάγερ, ότι στο Συμβούλιο και στα κράτη-μέλη χρειάζεται να πείσουμε για την κλίδα ε, κατανομής ε, στα πλαίσια του προϋπολογισμού. Και σας καλώ να ε, ε, πάρετε να ε, τα πείτε αυτά στα κράτη-μέλη, να προσπαθήσετε να τους νουθετήσετε για να το καταλάβουν. Ξέρω ότι δεν είναι δική σας δουλειά, αλλά τα κράτη-μέλη θα πρέπει να πιστούν. Συμφωνώ με την Άννα. Στη Γαλλία είχαμε πολύ θετικές εμπειρίες, ακριβώς σε μικρά χωριά. Οτιδήποτε έχει να κάνει με περιφερειακή συνεργασία, για να μην πω δημοτική συνεργασία ε, και κοινοτική σε επίπεδο δήμων και κοινοτήτων, δηλαδή βοηθάει. Διότι ε, όταν έχεις τα απόλυτα αριθμητικά στοιχεία είναι δύσκολο να καταλαβαίνεις περί τίνος πρόκειται. Ε, αλλά όταν βλέπει ο άλλος τι λειτουργεί στη πράξη και τι αποδίδει, προχωρούν τα ζητήματα που αυτή τη στιγμή είναι σε πλήρη εμπλοκή. Η κυρία Βαλέρο. Øh, Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλά αυτά τα οποία μας είπατε. Είδαμε τις λύσεις που μας περιγράφετε. Πιστεύω βέβαια ότι λείπουν κάποια πράγματα από την όλη συζήτηση όπως είναι οι συνθήκες ε, φιλοξενίας υποδοχής. Έχουμε πρόσφυγες ε, ή του άσυλο. Τα άτομα αυτά θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν ε, τη χώρα. Δηλαδή να βασιζόμαστε στις προτιμήσεις, τις επιθυμίες τους. Δεν θα πρέπει να είναι και κατάλληλη συνθήκη, θα πρέπει να υπάρχουν όμως αυτές τις χώρες κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης. κυρία Κιέγγε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την έκθεση και πρέπει να πω ότι είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας παρουσιάσατε και για τη δική μας δουλειά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πολιτική στη Μεσόγειο και για μια γενικότερη προσέγγιση. Πράγματι. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένες προτάσεις και δικές σας προτάσεις θα μας είναι χρήσιμες. πάντοτε πρέπει να προωθούμε την ανταλλαγή καλών πρακτικών, να ενισχύουμε αυτή την ανταλλαγή, το είπατε και εσείς και νομίζω ότι η καλύτερη χρήση και αξιοποίηση των μέσων, των πόρων θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα της εφαρμής ακριβώς καλών πρακτικών επιτόπου και μπορεί να βοηθήσει να γίνουν οικονομίες επιτόπου. Και αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο, επαναλαμβάνω. Νομίζω ότι θα πρέπει τα κράτη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να μπορούν να βασιστούν στα μέτρα που προτείνετε εσείς. Ένα άλλο ζήτημα είναι οι μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα. Για να υπάρξει διαφάνεια και στη χρήση των κονδυλίων έτσι θα αποφύγουμε τα κονδύλια που προορίζονται για τους ε, μετανάστες ή τους πρόσφυγες να μπουν στις τσέπες τελικά άλλων. Οι οποίοι μετά θα τροφοδοτούν το λαϊκισμό ή θα χειραγωγούν. Ενώ οι δικαιούχοι δεν θα έχουν πάρει καν αυτά τα χρήματα για τα, τα οποία προορίζονται για αυτούς και ολοκληρώνω με ένα τελευταίο στοιχείο που είναι η αμοιβαία αναγνώριση των συστημάτων ασύλου. Είναι ένα θέμα που θα το τονίσουμε, θα συνεχίσουμε να επιμένουμε. Να κάνω κι εγώ δύο σχόλια για δύο θέματα που μου έκαναν εντύπωση. Δεν αναφέρεται πουθενά την μετεγκατάσταση, το resettlement. Αυτό μου έκανε εντύπωση γιατί το θεωρώ από τα πιο σημαντικά μέσα των νομίμων δυνατοτήτων που έχουμε να προτείνουμε σε πρόσφυγες να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το δεύτερο, αν δούμε λίγο τη σκοπιά των κρατών μελών. Πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη, γιατί το σύστημα του Δουβλίνου εν μέρη προσκρούει και σε αυτό και από την δηλαδη Δηλαδή, υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που έχουν ένα πολύ ανεπτυγμένο σύστημα χορήγησης ασύλου, ενώ κάποια άλλα ανύπαρκτο. Και εκεί βαίνουν, λοιπόν ζητήματα που ε, παίζουν μεγάλο ρόλο. Για να εκτιμήσουμε τη δυνατότητα απορρόφησης ή ένταξης και ενσωμάτωσης σε ένα κράτος μέλλον. Αυτά είναι τα δύο που με έκαναν εντύπωση. Θα ήθελα να σας ξαναδώσω το λόγο για σύντομη ε, δευτερολογία για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες εκθέσεις. Thank you Ευχαριστώ, ήταν πολύ χρήσιμες ε, οι παρατηρήσεις. Για τις καλές πρακτικές θα αφήσω την Μάντλη να μιλήσει για χρήση των πόρων. Και το θέμα της αμοιβίας αναγνώριση είναι σημαντικό. Για την επανεγκατάσταση ή την μετεγκατάσταση. Το συζητήσαμε και ε, όταν ε, εξετάσαμε τις θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους. Χορήγηση βίσας ε, θεώρησης δηλαδή για να έρθουν και να αιτηθούν άσυλο κάποια άτομα εντός ένωσης. Συνάδελφός μου, ναι, πράγματι, για την απροθυμία να δοθούν περισσότεροι πόροι. Αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, ανησυχεί και το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή, το οποίο μελετά τις πρόσφατες προτάσεις της Κομισιόν, ανακατανομή κτλ. Τον, τον άσυλο. Αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε εδώ είναι μια κρίσιμη πρόκληση. Υπάρχει μια τάση. Φαίνεται σαν να μην γίνεται αντιληπτό το είδος της πρόκλησης που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους ευθυντές άσυλ. Από νομικής και πρακτικής πλευράς η πρόκληση είναι συλλογική. δεν μπορούν τα κράτη-μέλη με μονομερείς ενέργειες να περιορίσουν κάπως τα πράγματα. Και αν το αντιληφθούμε όλοι, ίσως καταλάβουμε ότι μάλλον χρειάζεται να υπάρξει ανακατανομή των πόρων εκεί που χρειάζονται. Όχι απαραίτητα σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Βέβαια το βλέπουμε ότι κάπου φτάνουν πολλοί πρόσφυγες Είδαμε στη Βορειοδυτική Ένωση, είδαμε στη Γερμανία, ενώ χώρες της Ένωσης είδαμε και στη Γερμανία να φτάνουν αρκετοί πρόσφυγες. Και σίγουρα υπάρχει και το θέμα της λειτουργίας του κοινού συστήματος ασύλου. Υπάρχουν επίσης συστάσεις συγκεκριμένες για τα κέντρα κράτησης και τους ε, καταβλισμούς ε, και τι συνθήκες ε, πρέπει να πληρούν. Είχαμε και την αναδιατύπωση οδηγίας του 2013 για τα κέντρα αυτά που δίνει κάποιες οδηγίες και για το εθνικό επίπεδο αλλά και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν καλύτερα τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Υπάρχει το γραφείο στήριξης ασύλου, το ΕΑΣΟ που μπορεί να βοηθήσει. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης και ανάλυση της πρότασης της Κομισιόν ε, για ε, relocation, κατάσταση, από δηλαδή ένα κράτος μέλος σε κάποιο άλλο. Βέβαια θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η πρόθεση και η βούληση του ετούντος άσυλο. Είναι και θέμα των δικαιωμάτων, αλλά είναι και θέμα πρακτικής, ε, πραγματικότητας, γιατί μια από τις αποτυχίες του συστήματο του Δουβλίνου είναι ότι δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τι προθέσεις και τις επιθυμίες των ατόμων, με αποτέλεσμα πολλοί να προσπαθούν να ε, παρακάμψουν τον κανονισμό και πηγαίνουν αλλού να μετεγκατασταθούν, ενώ αυτό ήθελε να εμποδίσει ο κανονισμός του Δουβλίν. Η Ιταλική Προεδρία πέρυσι ε, έθεσε κάποια ζητήματα τα οποία βέβαια μπορεί να μην έγιναν ε, ε, να μην ακούστηκαν τόσο πολύ και εμεί θέλουμε να τεθεί και το τεχνικό ζήτημα, δηλαδή σε σχέση με την ΕΜΕΒΕ αναγνώριση δύο τεχνικές ε, νομικές οδούς ερευνούμε και θα δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τις δύο σας και με ευγενικό τρόπο θα σας παρακαλέσω να αποχωρήσετε ε, και θα ήθελα να καλωσορίσω ε, τους επόμενους Γκαρσία Ανδράδα και Φίλιπ Μπρέκα. Thank Um Σε αυτή τη μελέτη πρόκειται για τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες ε, για την μετανάστευση. Καταφθάνουν οι δύο εμπειρογνώμονες uh, 10 λεπτά έχετε και οι δύο. Καθίστε παρακαλώ για να μπορέσουμε μετά στη συνέχεια να κάνουμε ερωτήσεις. exactly the change of names. Could you please give me your real name because you are not Mr. De Bruyke, I was informed. huh? Martin. Ah, Mr. Martin, that's fine, I had... Α, ο κύριος Μάρτιν, γιατί έλεγε ο κύριος Δεμπρούκ εδώ και είπα και εγώ. Ε, με χαρά σας καλωσορίζω, κύριε Μάρτιν. Who wants to begin? I will. So, Ποιο θέλει να αρχίσει. Ε, κυρία, ευχαριστώ. Είναι πολύ μεγάλη τιμή η ευκαιρία που έχουμε να σας παρουσιάσουμε τη μελέτη μας που μας ανέθεσε η Επιτροπή Ελευθεριών και να σας μιλήσουμε εξ ονόματος της ομάδας των, ε, των ερευνητών σε συνεργασία λοιπόν με τις τρίτες χώρες για τη μετανάστευση. Είναι ένα δίκτυο για τη μετανάστευση ε, και ο καθηγητής Ντερίκερ, η καθηγήτρια Χριστίνα Ορτάσα, ο συνάδελφος Ιβάν Μαρτίν και εγώ έχουμε τα εξή στοιχεία στην μελέτη μας. Πρώτα, ε, θα σας πω ποιο είναι το πλαίσιο και μετά ε, οι πολιτικές και οι προκλήσεις που έχουν να κάνουν μια τη συνολική θεώρηση της μετανάστευσης και της μετακίνησης πληθυσμών. έχουμε ένα θέμα εξωτερικής ε, αρμοδιότητας, ε, ενδοθεσμική και εξωθεσμική συνεργασία και συντονισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά ε, έχουμε συνολική θεώρηση και επισκόπηση όλων των δυνατοτήτων που υπάρχουν στην Ένωση για τη μετανάστευση, το άσυλο, τα πολιτικά, τα οικονομικά, τα νομικά και τα χρηματοδοτικά μέσα. Μετά, ε, εξάγουμε κάποια διδάγματα από ε, κάποιες βέλτιες πρακτικές που μας εμπνέουν και μετά ε, κάνουμε μια αξιολόγηση του αντικτύπου της συνεργασίας αυτής και με ποιον τρόπο επηρεάζει. Τρεις είναι οι διαστάσεις, η ουσιαστική πρώτα διάσταση, ε, λειτουργική στη συνέχεια, τα υπέρτα κατά και οι συνέπειες των μέσων και τέλος που ε, επιδέχεται βελτίωση το σύστημα και ο θεσμικός συντονισμός. Και τελειώνει η μελέτη με την παρουσίαση σύντομων μελετών ε, περιπτώσεων για το Μαρόκο, την Τινησία και τη Μολδαβία. Θα θέλαμε λοιπόν να σας παρουσιάσουμε κάποια πρώτα ευρήματα. Εγώ θα επικεντρωθώ στα μέσα συνεργασίας, τα πολιτικά, τα νομικά και ε, τα ε, θεσμικά και ο συνάδελφος Ιβάν Μαρτίν θα επεκταθεί σε άλλα θέματα. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της παρουσίας θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα ειδικά ερωτήματα που λάβαμε πριν αρχίσει η ε, μελέτη μας. Λοιπόν, ποια είναι ε, τα συγκεκριμένα στη συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Τα έχουμε χωρίσει με βάση τη φύση τους πολιτικά μέτρα που έχουμε διμερείς διαλόγους, ε, διαλόγους για την κινητικότητα, μετά έχουμε νομικά μέσα, ρήτρες μετανάστευσης, λεγόμενες ε, συλλογικές, συνολικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης και σύνδεσης και ειδικέ συμφωνίες για τη μετανάστευση, για την επαναπροώθηση, για την άρση της υποχρέωσης θεώρησης κτλ. Συστήματα περιφερειακά για την προστασία και άλλα. Frontex ε, και εξωτερική δράση της ΕΑΣΟ που αρχίζει αυτό τον καιρό και αναδύεται γεωγραφικοί στόχοι, εφαρμογή μέτρων. Η μελέτη μας κάνει μια συγκριτική ανάλυση του περιεχομένου των προτεραιοτήτων και των εφαρμοστικών μέτρων των μέσων αυτών και κάνουμε μια συγκριτική αξιολόγηση σε σχέση με τους στόχους που είχαν οριστεί στην αρχή. Περιφερειακοί διάλογοι, διμερείς διάλογοι ε, και άλλα ε, είναι κάποια μέτρα τα οποία μπορούμε ταυτόχρονα να δούμε σε πολλούς πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας για την ε, προώθηση της κινητικότητας και την ε, οργάνωση της νόμιμης ε, μετανάστευσης μπορεί να είναι επιθυμία αλλά δεν υπάρχει συγκεκριμένο μέτρο και μέσο για την κινητικότητα των εργαζομένων. Δεύτερος ο πυλώνας είναι ο πιο ολοκληρωμένος, η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης με την επανεισδοχή και τη διαχείριση των συνόρων. Ναι, μην μιλάς τόσο αργά. Πολύ γρήγορα μιλάω, μου λέει ο κύριος Μαρτίν, βεβαίως. Yeah, yeah, yeah, I have understood just, sorry, <laughs> first time. So... Ζητώ συγγνώμη δεύτερος πυλώνας, λέω, είναι ο πιο ολοκληρωμένος με μια σαφή ε, εστίαση στις συμφωνίες επανεισδοχής και τη διαχείριση των συνόρων, Frontex, ε, διάφορες συμφωνίες, εταιρικές σχέσεις κτλ. Ο τρίτος και ο τέταρτος πυλώνας Λοιπόν, δεν δίνεται αρκετή λοιπόν σημασία στους στόχους, ε, μόνο σε συμφωνίες RDPP και σε κάποιες δραστηριότητες της ΕΑΣΟ εκτός από κάποια άλλα ευρύτερα εργαλεία. Το ίδιο ισχύει για το τέταρτο πυλώνα για τη διεθνή προστασία. Τώρα, ποια είναι η φύση και η χρειά των μέσων. Ε, τα ε, ολοκληρωμένα μέσα, τα ευρύτερα, ε, είναι πολιτικά ουδέτερα ε, στα κράτη-μέλη, ε, ενώ κάποια άλλα που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν συντρέχουσες αρμοδιότητες όπως είναι η επανεισδοχή ή αποκλειστικές αρμοδιότητες των κρατών μελών όπως είναι η θεώρηση. Καμιά φορά είναι νομικά δεσμευτικά και άλλοτε όχι αυτά τα διάφορα μέσα. Ε, είναι ε, το ήπιο δίκαιο σε συμφωνίες εταιρικής σχέσης, συνεργασίας. Στο ουσιαστικό δίκαιο. Έχουμε λοιπόν κοινά ευρήματα και διαπιστώνουμε ότι οι ουσιαστικοί στόχοι συμπίπτουν γιατί αντιστοιχούν σε πυλώνες. Οι περιφερειακοί διάλογοι μπορούν να χαρακτηριστούν ε, πλαίσια συνεργασίας επικαλυπτόμενα και για τις ανατολικές χώρες και για τις χώρες της Αφρικής. Τα μέσα, ας πούμε, αν δούμε για τη δημιουργία δυνατοτήτων για την προστασία των προσφύγων, είναι κάτι που αντιμετωπίζεται ταυτόχρονα με εταιρικέ σχέσεις κινητικότητας, με το διάλογο για τη μετανάστευση, με διάφορα περιφερειακά προγράμματα και ακόμα με διάλογο για την απελευθέρωση θεώρηση σε βαθμό που διαφέρει ως προς την επιτυχία, τους στόχους και τα μέσα και την αποτελεσματικότητα. Επίσης, είναι απρόθυμα τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν σε αυτά τα ε, μέσα και εργαλεία. Αυτό ισχύει για όλα τα μέσα συνεργασίας, τα περιφερειακά, τα διμερή και τα γενικότερα. Ε, καλύτερα να είχαμε πιο λίγα μέσα, αλλά πιο αποτελεσματικά θα ήταν ε, κάτι που θα έφερνε θέμενη αξία, αλλά αυτό δεν το βλέπουν όλοι με το ίδιο ε, μάτι. Υπάρχουν ε, ανταγωνιστικές στρατηγικές σε θέματα εσωτερικών και σε θέματα εξωτερικής δράσης. Δεν έχουν όλη την ίδια θεώρηση ανάλογα με τη σκοπιά του καθενός. Σε ό,τι αφορά τις εταιρικές σχέσεις για την κινητικότητα, τα μεμονωμένα κράτη-μέλη έχουν πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από ε, πολυμερή έργα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κοινοτικά κονδύλια ε, που να επικεντρώνονται μόνο σε πολυμερή έργα και σχέδια που να έχουν εξασφαλισμένη προστιθέμενη αξία όχι να συνενώνουν κάποια διμερή προγράμματα των κρατών μελών με μια τρίτη χώρα και να είναι απλώς το άθροισμα Η εφαρμογή φαίνεται ότι δεν είναι ισόρροπη. Ε, θα πρέπει τα βαθμολόγια, οι πίνακες επιδόσεων να ε, ενημερώνονται τακτικά για να βλέπουμε τα ουσιαστικά πραγματικά αποτελέσματα και να αυξάνονται οι προτάσεις για την ανάπτυξη και τη μετανάστευση. Θα πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι πόροι για να υπάρχουν ε, δυνατότητες κινητικότητας για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις και επίσης ποικίλει το ενδιαφέρον των ε, εταίρων. Δεν δείχνουν όλοι τον ίδιο ενθουσιασμό. Ε, δηλαδή καλύτερα να γίνεται ίσως διαβούλευση και όχι πάντα πραγματικές διαπραγματεύσεις. Και τελειώνω με τα προγράμματα ε, περιφερειακής προστασίας, πράγμα που ενδιαφέρει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. το πεδίο εφαρμογή είναι πάρα πολύ ευρύ και αυτό μας δυσκολεύει ε, στο, στη μελέτη αντικτύπου. Υπάρχει έλλειψη συμβιβασμού στην ε, διαχείριση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε κάποιες χώρες. Ε, δεν πιστεύουν σε αυτά τα προγράμματα πάντα ε, όσοι τα χειρίζονται. Υπάρχει η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ που κάνει αντίστοιχες δράσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και χάνεται. Δεν προβάλλεται αρκετά η δράση της Ένωσης μέσα στο συνολικό πλαίσιο. Τα RPP, ε, η δράση είναι περιορισμένη. Τα κονδύλια μπορεί να έχουν αυξηθεί, να συμμετέχουν περισσότερο τα κράτη-μέλη από ό,τι στο παρελθόν Παραμένει όμως ε, μέγα το πρόβλημα στην προστασία των προσφύγων. Σε ό,τι αφορά το γκάμ που είναι η συνολική προσέγγιση στην κινητικότητα και στη μετανάστευση ε, χρειάζεται να δούμε πώς έχει σχεδιαστεί γιατί χωράει βελτίωση ε, θα πρέπει να επενδύουμε χρόνο και προσπάθειες για τη βελτίωση των μελετών αντικτύπου ε, για να δούμε κατά πόσο είναι αποτελεσματικές αυτές οι δράσεις και για τους εταίρους μας και για συγκεκριμένα πρόσωπα. Θα δώσω το λόγο τώρα στον συνάδελφο Ιβάν Μαρτίν για να μιλήσει για τη χρηματοδότηση. Ευχαριστώ πολύ, θα μιλήσω ισπανικά. Και με σεβασμό προς τους ε, διερμηνείς, σεβασμό για τους διερμηνείς σε ό,τι αφορά την εξωτερική συνεργασία στο άσυλο και τη μετανάστευση είναι μακρά η διαδικασία όπου η μετανάστευση και το άσυλο όλο και περισσότερο κυριαρχούν και αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο και σημασία στην εξωτερική συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναπτυξιακή συνεργασία αλλά και πιο πολιτική συνεργασία. Και ποιο είναι αυτό που έχουμε εδώ ως αποτέλεσμα. Ε, τέσσερις γενικές διευθύνσεις ή τέσσερις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής ασχολούνται πολύ ενεργά DEFCO, HOME, ε, NEAR και EAEV. Με πλήθος μέσων και εργαλείων για κάθε χώρα, για κάθε μεμονωμένη χώρα εταίρο που θέλει να συνεργαστεί για το άσυλο ή τη μετανάστευση. Για κάθε χώρα λοιπόν υπάρχουν 15 ή 16 διαφορετικά χρηματοδοτικά μέσα για να χρηματοδοτηθεί μία και μόνη δράση. Οπότε ποια ορατότητα. Καταλαβαίνετε ότι είναι περιορισμένη και πολλές φορές έχουμε επικαλύψεις. Για την προγραμματική περίοδο 2014 με 20 που διανύουμε, ο βασικό μέσο είναι το νέο θεματικό πρόγραμμα ε, δημοσία αγαθά και παγκόσμιες προκλήσεις για τη μετανάστευση και το άσυλο έχουμε 344 εκατομμύρια για μια πενταετία περίπου 50 το χρόνο είναι λίγο λιγότερο από ό,τι είχαμε στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο όλα τα υπόλοιπα κονδύλια που βλέπετε εδώ γεωγραφικά το μέσο συνεργασίας για την ανάπτυξη το Ταμείο για την μετανάστευση και διάφορα άλλα, για την εσωτερική ασφάλεια, ε, αστυνομία και σύνορα, το μέσο για τη γειτονία. Όλα αυτά λοιπόν δεν ξέρουμε πόσα χρήματα ε, πηγαίνουν από εκεί στη μετανάστευση. Δεν το γνωρίζουμε εκ των προτέρων, γιατί εξαρτάται από την υλοποίηση και την εκτέλεση. Για τα γεωγραφικά ταμεία π.χ. σε διμερές επίπεδο μόνο η Νιγηρία, Αιθιοπία και Μαρόκο έχουν θεωρήσει τη μετανάστευση προτεραιότητα στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά στα περιφερειακά προγράμματα είναι παρούσα η μετανάστευση. Πολύ σύντομα να δούμε πόση σημασία έχει εδώ η συνεργασία. Μόνο από την ΔΕΦΚΟ που είναι η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής Συνεργασίας έχουμε λεπτομέρειες μέχρι το 2013 αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς τι αφορά την εξωτερική συνεργασία. 100 εκατομμύρια το χρόνο είναι μέχρι το 2013, αυξήθηκαν λίγο τα κονδύλια, 45 με 55 εκατομμύρια ανάλογα με το έτος αφορούν τη μετανάστευση και το άσυλο και τώρα το τελευταίο πρόγραμμα τα δημόσια αγαθά και παγκόσμιες προκλήσεις και τα γεωγραφικά προγράμματα 2009 με 2011 αυξήθηκαν πολύ λόγω της διαχείρισης των συνόρων, της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων μετά από τις εταιρικέ σχέσεις για την μετανάστευση. Βλέπετε εδώ τις γεωγραφικές προτεραιότητες στην εξωτερική συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση. Βλέπετε τη γειτονία 20%, και το μοβ χρώμα είναι Ανατολική Ευρώπη. Το Μπορντό είναι η Βόρεια Αφρική. Ε, το Μπέζ εκεί είναι η ε, Ποσαχάρη Αφρική. Σε αυτές τις τρεις περιφέρειες αφιερώνεται το 60% περίπου τα δύο τρίτα ε, για τη συνεργασία στο άσυλο. Ενώ η Ασία και η Λατινική Αμερική κυρίως παίρνουν πολύ λίγα χρήματα. Ε, ε, ε, Και το τελευταίο slide τώρα διαφάνεια αυτή είναι η κατανομή των πόρων από το 2004 στο 2011 σε θεματικές προτεραιότητες. Ε, περίπου 30% έχει ως στόχο να ελέγξει την παράνομη μετανάστευση, 23% διεθνής προστασία και άσυλο, 24% ανάπτυξη και μετανάστευση που εκεί χωράνε πολλά πράγματα και μόλις 14% νόμιμη μετανάστευση και 10% δικαιώματα των μεταναστών. Αλλά εδώ θα πρέπει να πούμε ότι περιλαμβάνει εκστρατείες ενημέρωσης και εκπαίδευσης για την προστασία των δικαιωμάτων τους. Δεν, αφιερώνονται στην ίδια την προστασία των μεταναστών. Αυτά. Τελειώνω εδώ. Στα πλαίσια της μελέτης προσπαθούμε ε, να ε, συνδυάσουμε αυτά τα στοιχεία με εκείνα της Γενικής Διεύθυνσης ΚΟΜ επικοινωνίας δεν έχουμε πολλές φορές τα απαραίτητα στοιχεία στη διάθεσή μας για να κάνουμε την ανάλυσή μας, ενώ στην ε, αναπτυξιακή βοήθεια τα είχαμε στην DG DEFCO. Ευχαριστώ πολύ καταρχάς και τους δυο σας για τις παρουσιάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Η δική μου εμπειρία όταν διορίστηκα γενική συγγήτρια για τη Λιβύα επί Καντάφη δηλαδή για το τι προσέγγιση είχε η Ένωση ε, κατά τη διαπραγμάτευση συμφωνιών πλαισίου, όλα εξαρτώταν από τη Συμφωνία Επανεισδοχής. Και δεν ήταν κατανοητό αυτό που διακυβευόταν από πολιτικής πλευράς. εκ μέρους των κρατών μελών. Ήταν εξόφελμο. Ούτε καταλάβαιναν. Γιατί συνομιλούσαμε με το καθεστώς Καντάφη που είχε μόλις διώξει την υπατιαρμοστία, αρμοστία, είχε κακομεταχειριστεί με το στο δυνατό τρόπο τους μετανάστες. Δεν είναι καινούργια αυτά που βλέπουμε και επί αυτά τα γίνονταν. Mm. Άρα πραγματικά ήταν σοκαριστική έλλειψη αρχών. Και δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει και τίποτα ουσιαστικό. Βλέπουμε την ίδια έλλειψη αρχών να εκδηλώνεται με την απροθυμία φιλοξενίας ε, των ε, ενδεών αυτών ε, συμπολιτών, συνανθρώπων μας που ζητούν άσυλο. Ποιες είναι οι νομικές οδοί. Τα κράτη-μέλη εξετάζουν αυτό το ενδεχόμενο. Υπάρχει κάποιο κράτος μας που να έχει κάποιους νόμιμους διάβλους για τη μετανάστευση. Πώς έχουν τα πράγματα για αυτές τις νομικές οδούς οι νόμιμες. Είχα κι εγώ μια ερώτηση, αλλά πρώτα η κυρία Κιέγκε. Ε, Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και εγώ τους συντάκτες της μελέτης αυτής για τις παρουσιάσεις τους. Νομίζω ότι ακόμα πρέπει να γίνει πολλή δουλειά όμως, γιατί επί του παρόντος δεν είναι σαφής η σχέση ανάμεσα στη μετανάστευση, το άσυλο και τη διεθνή συνεργασία. Αυτό ήδη το βλέπουμε σε επίπεδο κρατών μελών, όπου τα Υπουργεία Εστερικών και τα Υπουργεία Εξωτερικών που είναι αρμόδια για τη συνεργασία δεν συνεργάζονται μεταξύ τους. Παρουσιάζουν εντελώς διαφορετικά και αποκλίνοντα προγράμματα και πραγματικά δεν ξέρω πώς θα καταφέρουμε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα να το εντάξουμε στις αρμοδιότητες ενός άλλου Υπουργείου όταν τα Υπουργεία Εσωτερικών και Εξωτερικών στα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συνεργάζονται επαρκώς. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο θέλω να θίξω είναι αυτό που έχει να κάνει με τους νέους. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα των νέων για τη διεθνή συνεργασία. Πρέπει να εργαστούμε πολύ και κυρίως για να ασχοληθούμε με τις νόμιμες οδούς της μετανάστευσης, αλλά πρέπει να δούμε και ποιες δυνατότητες έχουν ορισμένοι άνθρωποι προκειμένου να αναπτυχθούν, να εξελιχθούν στην ίδια τους τη χώρα. Μέσω της διεθνούς συνεργασίας λοιπόν θα πρέπει να ωφελήσουμε τους ίδιους τους νέους που αποτελούν πολύ συχνά το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού των τρίτων χωρών, για παράδειγμα στην υποσαχάρια Αφρική. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ότι μέσω της διεθνούς συνεργασίας μπορούμε πραγματικά να αλλάξουμε τα κριτήρια, την πραγματικότητα, του στόχου των ανθρώπων αυτών, να καταφέρουμε να επενδύσουμε περισσότερο σε νέους επιχειρηματίες, προκειμένου να καταφέρουν αυτοί να δημιουργήσουν περισσότερες ικανότητες, να εξελιχθούν στην ίδια τους τη χώρα. Δεν το κάνουμε όμως αυτό. Βλέπουμε ότι ε, στα σκάφη τα οποία έρχονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν κυρίως νέοι, άρα κάτι δεν πάει καλά. Εφόσον λοιπόν έχουμε κάποια μέσα στη διάθεσή μας, θα πρέπει να τα προσαρμόσουμε στην υφιστάμενη κατάσταση, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι οι οποίοι προσπαθούν να φύγουν από τη χώρα τους. Πώς μπορούμε να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους περισσότερες ευκαιρίες στην ίδια τη χώρα τους όμως, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε καλύτερη διακυβέρνηση, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ζουν σε, σε καθεστώτα δικτατορικά. Νομίζω λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να στηρίξουμε και με μία νέα κοινωνική τάξη στις χώρες αυτές μέσω των πόρων και μέσω των ε, εργαλείων αυτών που έχουμε ήδη στη διαθεσή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι μπορούμε λοιπόν εμείς να κάνουμε προκειμένου να έχουμε μια σφαιρική πολιτική, να συνδυάσουμε περισσότερο την εσωτερική με την εξωτερική μας πολιτική όταν αντιμετωπίζουμε τρίτες χώρες. Και όσον αφορά την εξωτερική αλληλεγγύη, νομίζω ότι και εκεί θα πρέπει να δούμε τους πραγματικούς λόγους της κρίσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ τους δύο επόμενους συναδέλφους να είστε σύντομοι, γιατί έχουμε άλλη μία μελέτη και δεν θα προλάβουμε να τους ακούσουμε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Έχω μια ερώτηση για το Μαρόκο και τα κονδύλια για το Μαρόκο. Τι εγγύησεις έχουμε ότι τα κονδύλια αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση του τείχους ε, στα κατεχόμενα εδάφη. <clears throat> Έχω και εγώ μια ερώτηση. Ακούσαμε πολλά για την οικονομική πτυχή. Εγώ θέλω να ρωτήσω για τις πρακτικές πτυχές της μετανάστευσης. Μιλάμε για τρίτες χώρες, πηγές, ε, οι χώρες προέλευση μεταναστών ε, ή μεταξύ τρίτων χωρών, από Αφρική προς ε, Σαουδική Αραβία, συνεργασία με την Αιθιοπία. Η συνεργασία έχει να κάνει με χριστιανούς, μετανάστες από την Ερυθρέα για παράδειγμα και τι γίνεται ακριβώς. Επίσης, θα ήθελα παραπάνω πληροφορίες για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στην πράξη τους πρόσφυγες στις τρίτες χώρες. Ich Τελειώνω εγώ και ε, σημειώνω αυτό που είπε είπατε εκπρόσωπο, κάποτε και πολύ σωστά ότι στην Αφρική δεν υπάρχουν μόνο φτωχές χώρες αλλά πάρα πολλές πλούσιες χώρες και η μετεκατάσταση ε, τους αφορά. Είναι 52 εκατομμύρια οι πρόσφυγες στον κόσμο. 52 εκατομμύρια. Και αυτοί δεν θέλουν να έρθουν μόνο στην Ευρώπη, δεν πρέπει να έρθουν μόνο στην Ευρώπη. Τι γίνεται με την ε, μετεκατάστασή τους στην Αφρική, ε, λόγω και του μεγέθους των καταστροφών και των ολέθρων, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρα από την ίδια συνεισφορά μας και υποδοχή στους ανθρώπους που ξεφεύγουν, από καταστάσεις που πρέπει να φύγουν να τους δώσουμε μια πατρίδα. Okay. Uh, Πολύ γρήγορα. Καταρχάς, η μελέτη αυτή είναι σε εξέλιξη. Σήμερα λοιπόν, πριν έρθουμε εδώ, συζητούσαμε ακριβώς με κάποιους από τους συναδέλφους σας το ζήτημα του πώς μπορούμε να εγγυηθούμε τον καλύτερο θεσμικό συντονισμό για τη συνεργασία στα πλαίσια της μετανάστευσης ε, και με την Κομισιόν και εντός της Κομισιόν. Ιδίω ε, τη ΓΔΧ και ΓΔΔΕΦΚΟ που φαίνεται να ακολουθούν όπως φαίνεται και επιτόπου διαφορετική λογική. Και θα έχουμε πολλά να πούμε στη μελέτη. Η πρόκληση σίγουρα έγκυται στο πώς μπορούμε να καταστήσουμε συμβατούς ε, δύο στόχους διαφορετικούς. Την εγκατάσταση χώρες προορισμού και την εκπλήρωση των στόχων της μεταναστευτικής πολιτικής της Ένωσης. Ό,τι αφορά τους νέους, οι μετανάστες κατά ποσοστό 80% είναι μεταξύ 18 και 30 ετών. Άρα προφανώς πρόκειται για μια πολύ σημαντική ομάδα στόχο θεωρώ ότι ένα πρακτικό ζήτημα αποκαλυπτικό, άκρος αποκαλυπτικό, είναι ότι το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση δεν υπάρχει σε αυτό ένα πυλώνας για την μετανάστευση και το άσυλο το αντιμετωπίζει ε, το θέμα της μετανάστευσης ως ένα θέμα που πρέπει να το διαχειριστούμε από την Ευρώπη. Κάποιες μικροαναφορές γίνονται στην νόμιμη μετανάστευση για τις παγκόσμιες ανισότητες ε, και το πλαίσιο της ανάπτυξης που σχετίζεται άρρηκτα με τη μετανάστευση. Για το Μαρόκο, ο βασικός κίνδυνος ε, ε, εκτροπής κάποιων κονδυλίων ή υπεξαίρεση κονδυλίων θα μπορούσε να γίνει στην περίπτωση της μεσονική στήριξης. Για την Ουκρανία και το Μαρόκο είναι οι δύο μόνες χώρες που στο παρελθόν Είχαμε προγράμματα δημοσιονομικής στήριξης για τη μετανάστευση περιορισμένα μεν, διακόπηκαν, δεν έχουν επαναληφθεί. Σήμερα λοιπόν ο κίνδυνος Ακόμη και τα προγράμματα ελέγχου συνόρων που χρηματοδοτεί η Ένωση, ε, για το Μαρόκο πάντα μιλάω, να χρηματοδοτήσουν τον έλεγχο συνόρων στη Δυτική Σαχάρα, αυτό το τείχος, είναι ε, κάτι που δεν μπορεί να υπάρξει ω κίνδυνο τεχνικά. Συνέβη κατά το παρελθόν, σήμερα δεν είναι πλέον δυνατόν. Για τι δύο τελευταίε ερωτήσει ε, μετανάστευση προ τον Νότο, Αιθιοπία, εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε ένα καλό παράδειγμα πριν από ένα χρόνο και δύο μήνε ακριβώ όταν η Σαουδική Αραβία 100.000 Αιθίωπες ή 110.000 Αιθίωπες ε, τους γύρισε πίσω και ήμασταν οι μόνοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ο μόνος χρηματοδότης που κινητοποιήθηκε για να βοηθήσει τα 110.000 αυτά άτομα και να τους δώσει προοπτικές στην Αιθιοπία, στο μέτρο του δυνατού πάντα. Και στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας ε, ε, γίνεται όλο και περισσότερος λόγος για την ανάγκη να έχουμε συνεργασία όχι μόνο τις ρο, προς το βορρά, νότος βορράς δηλαδή προς τη Βορευρώπη, αλλά να διαχειριστούμε καλύτερα και τις ροές από νότον προς νότον. Θα ήταν πολύ ε, σοβαρό σφάλμα να μην ασχοληθούμε και στο θέμα, με το, θέμα, για το θέμα αυτό και στη, στο θεματολόγιο για τη μετανάστευση και για τις πιο πλώσιες αφρικανικές χώρες. Οι πιο πολλές είναι χώρες ε, προ, ενώ Νότια Αφρική, Νιγηρία, Αλγερία. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει σίγουρα η πολιτική βούληση από πλευράς αυτών των χωρών για να λύσουν, για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσφέρει ένα συνολικό πακέτο ελκυστικό για να ασχοληθούν και αυτές οι χώρες. Όταν επιμείναμε όπως με το Μαρόκο, ενέκρινε νέο νόμο για το άσυλο νέα πολιτική μετανάστευση που είναι μοντέλο για την περιοχή. Άρα προς το παρόν, από τη μια λύπη ε, η πολιτική βούληση μεταξύ εντό αγωγικών πιο πλούσιες χώρες τη Βορειοαφρική, αλλά και η Ένωση δεν έχει ακόμη προσφέρει ένα ελκυστικό συνολικό πακέτο που να περιλαμβάνει και τα ζητήματα της υποδοχής προσφύγων, για παράδειγμα. Για ένα λεπτό, αν μου επιτρέπετε να κάνω δύο σχόλια, απαντώντα σε κάποια από τα ερωτήματα. Σε ό,τι αφορά την έλλειψη κατανόηση πολιτικής κατάστασης, την οποία μιλήσατε. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με αυτό που είπε και ο συνάδελφο: ότι απαιτείται και εσωτερικό συντονισμό εντός Επιτροπής, αλλά υπάρχουν και προκλήσεις. Συντονισμό μεταξύ ΕΕ και Κομισιόν, για παράδειγμα. Και το ρόλο των ε, αντιπροσωπιών της Ένωσης στις τρίτες χώρες πρέπει να δούμε υπήρξαν σύνδεσμοι που ε, πήγαν, ξανά πήγαν σε κάποιες χώρες τρίτες για να συζητήσουμε τα θέματα μετανάστευσης. Εκεί νομίζω είναι το κλειδί, αλλά το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει ένα είδος ανταγωνισμού για το ποιος έχει την τεχνική εμπειρία, τεχνογνωσία και το πολιτικό όραμα για αυτή τη στρατηγική, αλλά νομίζω ότι και οι δύο πλευρές είναι απαραίτητες. Ό,τι αφορά νόμιμες οδούς για την προστασία όσων έρχονται από αυτές τις χώρες. Εξ όσων γνωρίζω όλα τα κράτη-μέλη προοδευτικά εγκατέλειψαν αυτά τα είδη προστασίας που είχαν σε ισχύ και η Ελβετία τροποποίησε τους νόμους της ε, για να μην περιουστούμε στην επικράτεια της Ένωσης Τα, συζητήθηκαν, ε, τα συζητήσαμε τα περί και στην προηγούμενη έκθεση. Είπατε επίσης για την ολοκληρωμένη πολιτική των διαφόρων υπουργείων. Τα μέσα αυτά, ΓΑΜ, θέλουν να εξασφαλίσουν έναν εσωτερικό συντονισμό. Εσωτερικός συντονισμός στην τρίτη χώρα ουσιαστικά εξασφαλίζεται με αυτή την, ε, με αυτό το μέσο για την κινητικότητα. Ελπίζω το ίδιο να συμβεί και στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός πληροφόρησης για το τι γίνεται διμερός από τα κράτη-μέλη. Ακόμη και αν είναι εθνική αρμοδιότητα το θέμα. Έχουμε την αρχή της ε, συνεργασίας και επαναλαμβάνω θέλουμε συντονισμό και μεταξύ των Υπουργείων του ίδιου κράτους μέλους. Σταματώ εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε και άλλη μελέτη, ξέρετε. Έχουμε και άλλη παρουσίαση από πλευράς του κυρίου Μαρτίν και αν δεν το κάνουμε τα επόμενα δέκα λεπτά θα το χάσουμε για πάντα. Γιατί θα μας φύγουν οι διερμηνείς. so, Ευχαριστώ πάρα πολύ και να πάτε στο καλό. Έχετε το λόγο κύριε Μαρτίν μου. Θα είμαι πολύ σύντομος. Βλέπετε ότι έχει οριστικοποιηθεί σχεδόν η μελέτη, θα ολοκληρωθεί στο τέλος του μήνα. Πρόκειται για μια μελέτη που ζητήθηκε από το Migration Policy Center όπου εργάζομαι. Προσπαθούμε εδώ πέρα να εμπλέξουμε και ε, δικηγόρους και ειδικού ε, σε ζητήματα δημογραφίας και θέλουμε ουσιαστικά να δώσουμε μια πραγματική ουσία σε αυτή τη σφαιρική προσέγγιση στη μετανάστευση που αναφέραμε πριν από λίγο και θέλουμε να εστιαστούμε σε κάποιες νέες οδούς νόμιμης μετανάστευσης. Και έτσι απαντώ και στο ερώτημά σας. Ξέρετε ότι στην Ευρώπη υπάρχει το εξής παράδοξο. Χρειαζόμαστε οικονομικούς μετανάστες, αλλά από την άλλη δεν έχουμε τις νόμιμες οδούς για να τους φέρουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είμαι λοιπόν πολύ σύντομος. Βλέπετε εδώ πέρα τη διάρθρωση, τη δομή της μελέτης στην παρούσα της μορφή έχουμε έξι κεφάλαια όπου απαντάμε έξι ερωτήσεις. Θα κάνω ένα σύντομο σχόλιο για κάθε ερώτηση. Θα είμαι πολύ σύντομος λοιπόν καταρχάς. Για ποιο λόγο υπάρχει ανάγκη κοινοτική νομοθεσίας όσον αφορά την επαγγελματική μετανάστευση. Ουσιαστικά χρειαζόμαστε τέτοια νομοθεσία εξαιτία και τη ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να έχουμε ελεύθερη κυκλοφορία χωρί να έχουμε κοινή εργασιακή νομοθεσία, χωρί να έχουμε κοινή αγορά εργασία και χωρί να έχουμε κοινή πολιτική μετανάστευση στον επαγγελματικό τομέα. Απουσία τέτοια νομοθεσία υπάρχουν πάρα πολλέ δυσλειτουργίε στα πλαίσια τη ενιαία αγορά εργασία. Δεύτερον, Ποιε είναι οι ελλείψει που έχουμε εντοπίσει στην αγορά εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιε είναι οι προβλέψει όσον αφορά την μελλοντική επαγγελματική μετανάστευση. Εμεί ε, εξετάσαμε όλη την υφιστάμενη βιβλιογραφία και όλε τι εκθέσει και είδαμε ότι όντω η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη σήμερα χρειάζεται περισσότερου οικονομικού μετανάστε και πάλι Αντίθετα από ό,τι θα περίμενε κανείς, έχουμε περισσότερη ανάγκη σε μετανάστες με χαμηλότερες σχετικά επαγγελματικέ δεξιότητες και όχι ιδιαίτερα υψηλές επαγγελματικέ δεξιότητες. Και βλέπουμε, εστιαζόμαστε σε κάποιες χώρες όπως η Αυστρία, η Γερμανία και άλλες πλούσιες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντοπίσει 20 περιπτώσεις ε, αναγκών όσον αφορά την ε, επαγγελματική μετανάστευση και ουσιαστικά μόνο σε 8, 8 περιπτώσεις χρειαζόμαστε υψηλά εξειδικευμένους, ιδιαίτερα εξειδικευμένους μετανάστες. Φαίνεται ότι χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερους ε, μετανάστες μεσαίας ή χαμηλής εξειδίκευσης. Έπειτα, ποιο είναι το νομικό πλαίσιο όσον αφορά την επαγγελματική μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ μεγάλο εδώ κατακαιρματισμό, ανακατηγορία, χρειαζόμαστε ε, εξειδικευμένου ε, μετανάστες όσον αφορά την έρευνα, γίνεται αναφορά εδώ πέρα στην μπλε κάρτα, γίνεται αναφορά επίσης στους εποχιακούς εργαζόμενου, αλλά επίση και στου φοιτητέ. Υπάρχουν διαφορετικά μέσα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται όμω πολύ. Σε όλες τις μελέτες για την υλοποίηση και την εφαρμογή βλέπουμε ότι τα μέσα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή ανά χώρα δεν τα αποκρίνονται στις ανάγκες επαγγελματικής μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό αιτιολογείται από το ότι ε, αφήνεται πάλι μια πολύ μεγάλη διακρατική ευχέρεια στα κράτη-μέλη προς την εφαρμογή των μέσων αυτών. Επομένως, η δική μας προσέγγιση θα ήταν σε κεντρικό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή να δημιουργήσει μια σφαιρική προσέγγιση όσον αφορά την επαγγελματική μετανάστευση. Το τέταρτο τώρα κεφάλαιο έχει να κάνει με τον αντίκτυπο αυτών των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ μικρός αντίκτυπος γιατί υπάρχει όπως σας είπα πολύ μεγάλος κατακαιρματισμός, μικρή χρήση νηφιστάμενων εργαλείων, ωστόσο ένα κεντρικό ζήτημα που εντοπίσαμε είναι ότι οι πολιτικές αυτές δεν ενσωματώνουν αρκετά τους μη οικονομικούς μετανάστες που βρίσκονται ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα οι φοιτητέ, αυτοί που υποφελούνται του συστήματο επανένωση οικογενειών, δεν ενσωματώνουν του ετούντε άσυλο, οι οποίοι θα μπορούσαν να ενταχθούν, να ενσωματωθούν στην αγορά εργασία και να συμβάλλουν για να καλύψουν τι επαγγελματικέ ανάγκε στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν είχαμε κάτι τέτοιο, θα είχαμε και αυτό το οποίο ονομάζουμε σφαιρική προσέγγιση στην επαγγελματική μετανάστευση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέμπτον, το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση ανταποκρίνεται στι πραγματικέ ανάγκε Ευρωπαϊκή Ένωση για την επαγγελματική μετανάστευση. Η απάντηση είναι αρνητική. Δεν ανταποκρινόμαστε στα βασικά ζητήματα που έχουμε εντοπίσει, πώς θα μπορούσαμε δηλαδή να συνδυάσουμε τις ε, ανάγκες που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με, την, ε, με τις μεταναστευτικές ζωές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε μία μακροπρόθεση μόνο προσέγγιση με ένα σύστημα που χρησιμοποιεί πόντους, μόρια και θεωρούμε ότι το σύστημα αυτό δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες αγοράς εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες που έχουμε εντοπίσει. Το λέμε αυτό ξεκάθαρα στη μελέτη και το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Μετανάστευση θα μπορούσε να αποτελέσει χρυσή ευκαιρία για να αναλύσουμε και να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Το έκτο και τελευταίο κεφάλαιο της μελέτης προσπαθεί να εντοπίσει 18 διαφορετικούς νέους τρόπους νόμης μετανάστευσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και για κάθε από αυτές τις νόμες οδούς ζυγίζουμε τα θετικά και τα αρνητικά και αν πραγματικά ανταποκρίνονται στις ανάγκες αγοράς εργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλουμε να δούμε επίσης και το επίπεδο σκοπιμότητας σε πολιτικό-οικονομικό επίπεδο. Αναφερόμαστε στο πώς μπορούν να λειτουργήσουν αυτές οι νόμιμες ε, οδοί, αντιστοίχηση πραγματικών αναγκών και οικονομικών μεταναστών, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να καλύψουμε τις οικονομικές ανάγκες Ευρωπαϊκής Ένωσης τους ήδη υφιστάμενους μετανάστες, φοιτητές, όσους έχουν επωφεληθεί από τα συστήματα οικογενικής επανένωσης. Κάνουμε επίσης μια διασύνδεση εδώ πέρα με προηγούμενες μελέτες. Θέλουμε να συνδυάσουμε τις ανάγκες αυτές της επαγγελματική μετανάστευσης με άλλες πολιτικές όπως η πολιτική γειτονίας και αναθεωρούμε κάποιες ε, υποχρεώσεις όσον αφορά το σύστημα αναφοράς, το σύστημα δικτών που χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη. Δυστυχώς δεν υπάρχει συστηματική παρακολούθηση της εθνικής πολιτικής μετανάστευσης των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει απαραίτητη διάρθρωση δηλαδή και ζητάμε επίση και περισσότερη διαβούλευση με όλου του εμπλεκομένου. Ευχαριστώ. Εγώ σα ευχαριστώ. Μία ερώτηση, αν θέλετε, τώρα όμως και πολύ σύντομα για να τελειώνουμε. Κύριος Γιούρεκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα κάποια σχόλια θέλω να κάνω. Για τι πράγμα μιλάμε εδώ. Πριν από πέντε χρόνια μια μεγάλη ομάδα κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιόριζε τη δυνατότητα άλλων Ευρωπαίων πολιτών να εργάζονται νόμιμα ε, στην επικράτειά τους. Έχουμε μεγάλες ροές μεταναστευτικές, εσωτερικές, εκτός από τις εξωτερικές. 500.000 ανέφερε ε, η κυρία Γκόμες στις Πορτογάλους που μετανάστευσαν, που ξενιτεύτηκαν. Κοιτάξτε τι γίνεται. Πάνω από το 10% των πολιτών της Βουλγαρίας, ε, Φερρυπίν, ή της Λιθουανίας μετακινούνται και ε, προκαλούν τεράστιες ε, αντιδράσεις ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για να μην μιλήσω για τους πολίτες της Ένωσης που κυκλοφορούν. Αυτό πώς το συγκρίνεται με την εξωτερική μετανάστευση. Εδώ μπλοκάρεται η αλληλεγγύη προς τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανθρωπιστική βοήθεια είναι άλλο πράγμα και άλλο η μετανάστευση. Η Άννα, πολύ σύντομα για να βάλουμε στο πλαίσιο τις 485.000 Πορτογάλους που έφυγαν. Οι περισσότεροι έχουν προσόντα και δεξιότητες και δεν μπαίνουν στην ίδια κατηγορία των οικονομικών μεταναστών. Είναι απόδημοι, expatriates, δεν είναι οικονομικοί μετανάστες. because of the crisis. Έχουν φύγει γιατί δεν βρίσκουν δουλειά στη χώρα τους. Δεν είναι οικονομικοί μετανάστες. Θα προτιμούσαν να είχαν βρει δουλειά στην Πορτογαλία. Σας διαβεβαιώ. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και μετανάστευση εκτός από χώρα ε, προέλευσης που όψιμοι είμαστε ε, έχουμε και ε, υποδοχή μεταναστών από τη Μολδαβία, την Ουκρανία, την Αφρική, τη Βραζιλία που είχαμε μετανάστες στο παρελθόν. Ήμασταν χώρα προορισμού. Βέβαια ήταν οι πρώτοι που έφυγαν με την ε, μετανάστευση. Αλλά τώρα πάσχουμε γιατί έχει αποψηλωθεί η ύπεθρος και χρειαζόμαστε επιγόντως ανθρώπους, ε, μετανάστες. Είναι γελίο που δεν το καταλαβαίνουν οι κυβερνήσεις. Ε, γιατί δεν, δεν το καταλαβαίνουν και αν το καταλαβαίνουν δεν θέλουν να το κάνουν νόμιμο, δυνατό και ασφαλές αυτό. Μια σύντομη παρατήρηση στο Ηνωμένο Βασίλειο ζητούσαν διακαώς νοσηλεύτριες από την Πορτογαλία και το ξέρω εξαιτίας πείρας διότι ήταν εξαιρετικέ και στην εκπαίδευση και γενικότερα. Τρία πολύ γρήγορα σχόλια. Όταν μιλάμε για νόμη μετανάστευση και για αυτή μιλάμε στην έκθεση, μιλάμε για τις χώρες. Ε, το ίδιο συμφέρον των χωρών της Ένωσης. Δεν μιλάμε ούτε για αλληλεγγύη ούτε για συνεργασία. Μιλάμε για κάλυψη των αναγκών της Ευρωπαϊκής Αγοράς Εργασίας πρώτον. Δεύτερον, προφανώς είναι και πολύ λεπτό από πολιτική πλευρά το ζήτημα. Το γνωρίζουμε όλοι. Δική μας υποχρέωση ως ακαδημαϊκών και ερευνητών είναι να σιγουρευτούμε ότι συλλέγονται οι σωστές πληροφορίες και διαβιβάζονται και αυτές οι πληροφορίες είναι η βάση γιατί ο σχηματισμό πολιτικών δεν γίνεται πάντα αυτό μέχρι τώρα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν για να απαντήσω και με αυτό τελειώνω στο ερώτημά σας, ε, για να απαντήσω λοιπόν, τι μελέτη έχουμε τα εξή βασικά πορίσματα. Για να ε, έχουμε την εσωτερική κυκλοφορία των Ευρωπαίων πληθών θα πρέπει να τη συσχετίσουμε με την νόμιμη μετανάστευση, ε, την οικονομική μετανάστευση, που φαίνεται να είναι δύο διαφορετικά πράγματα από οικονομική πλευρά για του εργοδότε τη Ένωση, ε, για του Γερμανού για παράδειγμα εργοδότε. Το αν έρχεται ο εργαζόμενο από το Μαρόκο και την Πορτογαλία του είναι μια ή άλλη. Το θέμα είναι να είναι αποτελεσματικοί και να έχουν την νόμη δυνατότητα να εγκατασταθούν στη χώρα. Αυτή είναι, κατά την άποψή μου, η πρόκληση. Και αυτή είναι η βασική ε, εστίαση της οικονομικής μετανάστευσης. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Κερδίζετε το βραβείο ε, των ε, πιο ακριβέστερων και ταχύτερων πληροφοριών της ημέρας, αλλά ταλαιπωρείται τους διερμηνείς, οι οποίοι κερδίζουν και αυτοί το βραβείο της πιο γρήγορης ε, μετάφρασης της ημέρας. Πάμε στα διάφορα τώρα, δεν ξέρω αν έχει κανείς κανένα διάφορο, παραμονές καλοκαιριού, να πει τίποτα, τώρα να μιλήσει, τελείως να σοπάστε γιατί πάμε για καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι καλές διακοπές. Ελπίζω όλοι να επιστρέψετε την 3η του Σεπτέμβρη ξεκούραστοι και με χαρά να τα πούμε στις 9 η ώρα το πρωί. Σας εύχομαι να επανέλθετε με υγεία και ε, με ε, καλή διάθεση στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ πολύ.